Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώ ήρθατε στην Επιτροπή σε Περιβάλλοντος. Οι απογευματινές συνεδριάσεις ε, αργούν να αρχίσουν, ε, αργούν οι συνάδελφοι να έρθουν, αλλά σιγά σιγά θα γεμίσει η αίθουσα. Οι συντονιστές δεν χρειάζεται να συνεδριάσουν, αυτή είναι μια πρώτη ανακοίνωσή μου, τα είπαμε όλα και τα λύσαμε στο Στρασβούργο. Οπότε στις 6 δεν θα λάβει χώρα η συνάντηση, η συνεδρίαση των συντονιστών. Εστονία, Λετωνία, ε, εστονικά, λετωνικά δεν έχουμε και αύριο ε, μαλτέζικα δεν έχουμε. Επίσης ε, βλέπετε εδώ από το Ηνωμένο Βασίλειο ε, ένα κινηματογραφικό συνεργείο που θα ε, πάρει κάποιες λήψεις σχετικά με το ε, τρόπο των εργασιών μας. Δεν θα έχετε αντίρρηση ελπίζω. Η Europal TV αύριο θα παρευρεθεί για να κινηματογραφήσει την συνάντησή μας με τον πρόεδρο Μπούζεκ, περιβαλλοντικές προσπάθειες που κάνει το Κοινοβούλιο στα κτίρια του και στη λειτουργία του. Και έτσι περνάω στο σημείο 3. Α, στο 2 ακόμα. Δύο-τρεις ε, ανακοινώσεις από την προηγούμενη συνεδρίαση. Εδώ έχουμε μια, ένα καλό έργο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έναν ε, άτλαντα για την κατάσταση των εδαφών σε ορισμένα κράτη-μέλη. Υπάρχει στη γραμματεία για να το δείτε, ίσως και στο διαδίκτυο στο Ηνωμένο Βασίλειο, Μπενελούξ, Βόρεια Γαλλία, εδάφη ε, και περιοχές πυκνοκατοικημένες και υπάρχουν φόβοι για διάσπαση των εδαφών, αποδόμησή τους και η οδηγία για τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα μόνιμο θέμα στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής μας. Ένα άλλο μάλλον δυσάρεστο θέμα ο ΙΚΑΟ, ε, Διεθνής Οργανισμός για την Αεροπλοεία, συνεδριάζει αυτή την εβδομάδα στο Μοντρεάλ και ορισμένες ε, ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες προσέφυγαν κατά της εμπορίας εκπομπών στις αεροπορικές μεταφορές όπως είχε αποφασιστεί για το 2008. Την περασμένη εβδομάδα επ' αυτού ε, έλαβε χώρα μια αρκετά διεξοδική συνάντηση το βράδυ στο Στρασβούργο και ελπίζω η ΕΠΑ με τον Καναδά και το Μεξικό να μην καταφέρουν να περάσουν ένα ψήφισμα το οποίο θα συντρίψει την εμπορία των εκπομπών γιατί και η αεροπλοεία και η ναυσιπλοεία αποτελούν σημαντικά στηρίγματα στην μάχη μας για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτές τις μέρες αρχές της εβδομάδας ελάβαμε και μία ανακοίνωση της Κομισιόν για την οδηγία για τον καπνό. Επεξεργασία της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού. Υπάρχουν ορισμένα στο pipeline, ετοιμάζονται και έχει να κάνει και με ψηφίσματα για το κάπνισμα και την υγεία. Και οι συνάδελφοι μπορούν να μελετήσουν κάποια στιγμή σε βάθος τι προβλέπει η Κομισιόν στον τομέα αυτών. Στη Νέα Υόρκη, γύρω από το Σύνοδο Κορυφής της Χιλιετίας, έλαβαν χώρα και συνεδριάσεις για τη διάσκεψη για το κλίμα στο Κανκούν και μια υψηλού επίπεδου συνάντηση για τη διάσκεψη της βιοπικιλότητας στην Αγκόγια και ακούω ότι ο συνάδελφος Αρσένης παρευρέθη και ίσως έτσι κάπως συνοπτικά θα μπορέσει να μας ενημερώσει σχετικά με το αποτέλεσμα. Ίσως δεν έχουμε πολύ χρόνο βέβαια, αλλά κάποια πράγματα, έτσι λίγες ε, φράσεις θα μπορέσει να μας πει ο κύριος Αρσένης για την ε, βιοποικιλότητα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνάντηση και τις τέσσερις ημέρες που κράτησε. Η πρώτη μέρα αφορούσε την βιοπικιλότητα, ε, συζητήσεις υψηλού επίπεδου για τη βιοπικιλότητα το πρωί. Δύο θέματα που συζητήσαμε στην Επιτροπή μας επίσης συζητήθηκαν. Δεν θα υπάρξει συμφωνία στην Αγκόγια, εκτός και αν υπάρξει συμφωνία για τα γενετικά υλικά και υπάρξει συμφωνία για τη χρηματοδότηση. Αυτό το ξεκαθάρισαν όλοι οι ηγέτες των ε, αναπτυσσομένων χωρών. Η Βραζιλία ασχολείται με τα γεννητικά υλικά και εστιάζεται σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν ε, στέκεται στο πλευρό των αναπτυσσομένων χωρών. Εμείς μπλοκάρουμε τις συζητήσεις για ένα πιο φιλόδοξο πρωτόκολλο που θα εγγυάται ότι τα γενετικά υλικά που χρησιμοποιούμε και τα οποία προστατεύονται από διπλώματα ευρυσιτεχνίας παρόλα αυτά τα απελευθερώνουμε ούτως ώστε οι γηγενείς πληθυσμοί να μπορούν να υποφεληθούν και αυτοί από αυτά τα υλικά. Ευχαριστούμε πολύ για τη σύντομη αυτή ενημέρωση. Ε, διαμορφώνονται δύσκολα οι σχέσεις βορρά-νότου, φτωχών, πλούσιων και σε αυτό το θέμα. Θα δούμε τι εξελίξεις θα υπάρξουν ακόμη μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, περνάμε στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης για να εγκρίνουμε τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης του Ιουλίου. Μέχρι το τέλος της συνεδρίασης μπορούμε να δεχτούμε διορθώσεις. Αν δεν υπάρξουν θα θεωρηθούν εγκριθέντα. Και περνάμε στο κύριο θέμα της απογευματινής αυτής συνεδρίασης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να καλωσορίσω εδώ την Επίτροπο Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, η οποία είναι Επίτροπος για τη Διεθνή Συνεργασία, την Ανθρωπιστική Βοήθεια και την Αντιμετώπιση των Κρίσεων. Και αυτό το τελευταίο, αντιμετώπιση κρίσεων, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Και χαιρόμεθα πολύ που βρήκατε χρόνο, κυρία Επίτροπε, να έρθετε εδώ στην Επιτροπή πρόσφατα ή τον τελευταίο καιρό τέλος πάντων είδαμε μεγάλες καταστροφές και διεθνώς αυξήθηκαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Για να μην πω διπλασιάστηκαν υπάρχουν ξηρασίες αφενός και πλημμύρες από την άλλη. Επίσης ε, πυρκαγιές στα δάση και πολλά άλλα όλο και πιο ακραία φαινόμενα. Και οι πολίτες βέβαια αναρωτιόνται τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως ώστε να ε, αξιοποιήσει το δυναμικό που υπάρχει στην Ευρώπη, γιατί είμαστε μια ήπειρος με πολλές δυνατότητες αναξιοποίητες και πολλές φορές συζητήσαμε για το πώς θα δημιουργήσουμε συνέργειες μέσα από συνεργασίες και μέσα από ολοκληρωμένες ενέργειες, ούτως ώστε να πετύχουμε το καλύτερο για τον άνθρωπο και τη φύση. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε τι συζητείτε στη Νέα Επιτροπή, τι έχετε υπόψη σας να κάνετε σε επίπεδο νομοθεσίας, αλλά και σε επίπεδο προγραμμάτων και δραστηριοτήτων. Ένα θερμό καλώς ήλθατε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και σας δίνω το λόγο για την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι βουλευτές, είναι για μένα μεγάλη τιμή το ότι είχα την τύχη να βρεθώ σήμερα εδώ και ξέρετε η σταδιοδρομία μου όλη ήταν αφιερωμένη σε θέματα περιβάλλοντος. Οπότε και για αυτό νομίζω ότι θα μπορέσω να συνεισφέρω στον προβληματισμό σας. Σήμερα αυτό που θέλω να κάνουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ε, δυνατότητα αντίδρασης στις φυσικές καταστροφές, θεομηνίες κλπ. γι' αυτό το κοινοβούλιο απευθύνθηκε στην Επιτροπή αρχά του έτου και είπε ότι θέλει να υπάρχει ένα μηχανισμό ταχεία αντίδραση. Οπότε και εγώ αυτό που θέλω είναι να σα πω ποιε είναι οι προτάσει που ε, θα στοχεύουν στο να ανταποκριθούμε σε αυτό το οποίο θέλετε και να ανταποκριθούμε και εις τις απαιτήσει και προσδοκίες που υπάρχουν ε, διότι κύριε Πρόεδρε έχουμε όλο ένα και περισσότερες τέτοιες φυσικές καταστροφές και η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει από το 1975 έχουμε με πενταπλάσια συχνότητα τις θεομίες που συμβαίνουν βέβαια ε, ταυτόχρονα η οικονομία του πλανήτη έχει μεγαλώσει τρεις με τέσσερι φορέ και όμως βλέπουμε ότι οι θεομηνίε είναι πιο δυνατές από αυτή την οικονομική βελτίωση και έχουμε, και έχουμε καταγράψει κάποιες, ε, κάποια, κάποια εξαιρετικά φαινόμενα έχουμε τα 230 εκατομμύρια φέτος που έχουν πληγεί από τέτοιες καταστροφές και 85.000 έχουν ε, σκοτωθεί. Η δαπάνη είναι 66, 67 δις ευρώ. Η χρηματική αποτίμηση αυτών των καταστροφών. Φέτος πάντως δεν ήταν με τίποτα μία μέση χρονιά. Και θυμάμαι ένα καθηγητή που μου ε, έλεγε, που μου δίδασκε στα σχέδια ότι μπορεί κανεί να βάλει τα, τα, τα, πόδια στο φούρνο, το κεφάλι στην κατάψυξη και η, η μέση θερμοκρασία θα είναι ίδια, αλλά παρόλα αυτά θα πεθάνει. Βλέπετε μέσα ότι είχαμε αυτό το 2010 που ήταν χρονιά πραγματικά εξαιρετική, γιατί είχαμε την θεομηνία στην ΑΕΤ, όπου είχαμε 230.000 που πέθαναν 300.000 ε, περίπου τραυματίστηκαν, ένα εκατομμύριο μείναν οι Είχαμε την έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία, όπου επί έξι ημέρες ε, σταμάτησαν ενέργειε ε, μεταφορές, οι και είχαμε κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που ήταν κάτι το οποίο ξεπέρασε τα ευρωπαϊκά σύνορα. Επίσης είχαμε την έκρηξη, την υποθαλάσσια όπου σκοτώθηκαν κάποιοι 11 περίπου εργαζόμενοι και στον κόλπο του Μεξικού. Ε, επίσης είχαμε τέτοια φυσικά φαινόμενα που ακόμα δεν έχουμε καν αποτιμήσει τις συνέπειές τους. Και στην Ευρώπη είχαμε πλημμύρες, Ρουμανία, Μολδαβία, Σερβία, Ουκρανία. Παντού, παντού είχαμε πλημμύρες μέσα σε ένα και μόνο καλοκαίρι. Όμως από την άλλη μεριά στο Σαχέλ είχαμε ξηρασία και ελπίζουμε πάντως ότι εκεί κάτι θα κάνουμε ε, και δεν θα φτάσουμε σε φάση ε, ανθρωπιστικής καταστροφής όπως το 2005 και βλέπουμε μόνος ότι κάποια πράγματα είναι πέρα από δυνατότητες διαχείριση. Επίση, πλημμύρισε στο Πακιστάν. Οπότε θα πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση στη χώρα εκείνη με ανησυχεί πάρα πολύ, διότι διαπιστώθηκε ότι η τάξη μεγέθους ήταν ε, τρομερή. Μιλάμε για 20 εκατομμύρια ε, πληγέντων προσώπων στο Πακιστάν και βέβαια δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι πρόκειται τα πράγματα να είναι υπιότερα ή στο μέλλον. Αλλάζει το κλίμα. Έχουμε ένταση συγκέντρωση του πληθυσμού, αύξηση του πληθυσμού, κυρίως σε αστικές περιοχές και κατά τρίτο λόγο και αυτή και μόνη η, η ποικιλία και το βεληνικές της παγκόσμιας οικονομίας μας οδηγεί σε φαινόμενα σαν αυτό που είχαμε στον κόλπο του Μεξικού. Αλλά, οπότε και με όλα αυτά τα δεδομένα έχει καταστεί σαφέ ότι δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη ότι 90% των πολιτών απαιτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες της όσον αφορά την ε, αντίδραση σε αυτά τα φαινόμενα. Και ακριβώ αυτό δεν λέμε ότι πρέπει να κάνουμε. Κάνουμε κάτι όπω το παιδί. πραγματικότητα, όπω το ζητούν οι πολίτε. Για να δούμε επομένω τι μπορούμε να κάνουμε για να φέρουμε τη διαφορά. Γιατί έχουμε τέσσερι τομεί όπου είναι πάρα πολύ βασικό ότι να υπάρχει συντονισμό. Χωρί όμω να δυναμητίζουμε το ότι πρέπει να έχουμε ευθυγράμμιση, συντονισμό δυνατοτήτων, ευθυνών, και ε, να έχουμε αποκέντρωση. Δηλαδή τη βασική ευθύνη δεν έχει η τοπική κυβέρνηση, να τον έχουν οι τοπικέ αρχέ, να έχουν οι εθνικέ κυβερνήσει. Όμω είναι πολύ σημαντικό αυτό που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα-πρώτα. Όταν κάποια χώρα χτυπιέται από μια τέτοια θεομηνία, να έχουμε ένα σωστό συντονισμό, ούτω ώστε να μπορούμε να έχουμε όλα τα επιπλέον στοιχεία, όλη την εμπειρογνωμοσύνη που χρειάζεται για να μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συγκρατήσουμε το, το, το, το κόστο το οικονομικό και το κοινωνικό, γιατί χωρί το συντονισμό υπάρχει ο κίνδυνο που να έχουμε επικαλύψει, να έχουμε και αναποτελεσματικότητα. Δεύτερον, χρειάζεται να έχουμε κοινή εκπαίδευση και να αναδιδασκόμεθα από την εμπειρία, να αναβαθμίσουν τα εθνικά συστήματα, ούτως ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, υπάρχουν ε, κάποια μέσα που είναι στη διάθεσή μας που περισσότερο βοηθούν εις κοινωνικό επίπεδο. Είτε επειδή είναι πολύ δάπανα, είτε επειδή χρησιμοποιούνται πάρα πολύ σπάνια και επομένως δεν έχει νόημα η χώρα να, να αγοράσει αυτά τα μέσα. Ε, να επενδύσει σε αυτά. Τελευταίο όμω και σημαντικό ότι χρειάζεται μια συντονισμένη δυναμική αντίδραση Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα επίπεδα ώστε ε, να είναι και εικόνα που δίνουν προ τα έξω καλύτερη και ταυτόχρονα να ανανεώνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στο ότι μπορούμε κάτι να κάνουμε για να διαχειριστούμε ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο. Άρα, τι προτείνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε Ήδη σήμερα υπάρχει ένα σύστημα αντίδρασης. Είναι ικανοποιητικό. Όταν είχαμε τις πλημμύρε της Κεντρικής Ευρώπης, μέσα σε λίγες ώρες, κινητοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη όσα ζητήθηκαν και ακόμα περισσότερα. Όταν επίσης αντιδράσαμε ε, στις, πλημμύρε του Πακιστάν, ε, έγινε αυτό με συντονισμό των μελών, είχαμε και αέρια επέμβαση Ακριβώς αυτό το θεώρησαν πάρα πολύ θετικό οι αρχές του Πακιστάν και είχαμε 25 κράτη-μέλη που βοήθησαν την ΑΕΤ και αυτό έγινε αποτελεσματικά και συντονισμένα. Άρα εδώ δεν ξεκινούμε από το 0, από το α. Έχουμε κάποια πράγματα, κάποιε επιδόσει μας κάνουν περήφανος όμως. έχουμε ήδη αντλήσει κάποια μαθήματα από το ότι έχει γίνει στο παρελθόν, από όσα λέει η έκθεση Μπαρνιέ, με κατόπιν διαβουλεύσεων με τα κράτη-μέλη αλλά και από τα όσα μας έχουν πει και προτείνει όλοι οι εμπλεκόμενοι. Και έτσι λαμβάνουμε υπόψη όλα αυτά το μπορούμε να κάνουμε τα επικοινωνία στους αμέσους μήνες, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι βασικά το να απομακρυνθούμε από αυτό το οποίο σήμερα ισχύει, δηλαδή που είναι μια αντίδραση ad hoc. Δηλαδή γίνεται μια θεομηνία, κλίση και ανάπτυξη μέσων αντίδρασης. Άρα θα έχουμε τώρα ε, προπαρασκευή, ε, πρόβλεψη και άμεση ανάπτυξη μέσων αντίδρασης. Ε, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και προτείνουμε στα κείμενα ανακοινώσεων είναι πρώτα-πρώτα να προγραμματιστούμε βάσει κάποιων σενάριων τι θεομηνίε περιμένουμε να μα χτυπήσουν. Δεύτερον, να και να αποτιμήσουν τη μέσα έχουμε στη διάθεσή μα και επίση να προωθούμε στα κράτη-μέλη, ώστε σε εκούσια βάση να μα διαθέσουν ό,τι μέσα στη διάθεσή τους και επομένως όταν ε, καλώ κάποιο κράτος μέλος να μην αγωνιώ ποια θα είναι η απάντηση. Να ξέρω από πριν ποιος θα δώσει και τι και πόσα τέτοια μέσα για τη συγκεκριμένη φυσική καταστροφή, θεομηνία. Τρίτον, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν ρυθμίσεις ε, μεταφοράς πάνω σε αυτό το κοινοβούλιο ξεκαθάρισε τη θέση του, το τι περιμένει. Ε, επίσης, προτείνουμε και προβλέπουμε να έχουμε μεγαλύτερο συντονισμό ε, επιμελητίας όσον αφορά τις τρίτες χώρες όπως στην Αϊτή, όπως το Πακιστάν και έτσι με αυτή την επιμελητία να μπορούμε να έχουμε και ανάπτυξη κάποιων μέσων τα οποία θα συντεριάξουν με τα κοινοτικά και αυτά που κάνουμε από την Ένωση να έρχεται και να δένει με τα άλλα και έτσι να υπάρχει συντονισμό στην αντίδραση. Και έτσι θα έχουμε έναν πυρήνα ικανότητα αντίδραση τη Ένωση και για δράσει εκτό ΕΕ. Πρόκειται να συνεργαστούμε με την ε, κυρία Άστον, με την υπηρεσία εξωτερική δράση, ώστε να μπορούμε και εμεί να συνεισφέρουμε και να έχουμε μια συνολική αντίδραση τη Ευρώπη για τέτοιου είδου μεγάλες ε, καταστροφέ και θεομηνίε. και βεβαίω σε αυτές τις περιπτώσει θα πρέπει να έχουμε και ανάπτυξη στρατιωτικών μέσων ανάλογα με το τι απαιτούν οι περιστάσεις. Τελευταίο, στην ανακοίνωση τονίστηκε το πώς θα γνωστοποιήσουμε στον κόσμο αυτό το οποία κάνουμε γιατί πολύ συχνά απορεί ο κόσμος για το τι κάναμε, αν απέδωσε αυτό που κάναμε, αν ήταν σωστό αυτό που κάναμε. Έχουμε τώρα και άλλες προτεραιότητες σε σχέση με τις φυσικές καταστροφές βασική προτεραιότητα είναι το να υλοποιηθούν οι συστάσεις της ανακοίνωσης όσον αφορά την πρόληψη και την ετοιμότητα. Και σχετικά με αυτό σας λέω το ότι ήταν πάρα πολύ θετική η έκθεση Φερέιρα της Ολομέλειας του Σεπτεμβρίου. Και για να μπορέσει μια τέτοια προσέγγιση να αποδώσει θα πρέπει να έχουμε οριζόντιο συνδυασμό όλων όσων έχουμε στη διάθεσή μα. Την οδηγία του Σεβέζου, του, του, του, την άλλη για τι πλημμύρε και για την αποτίμηση των συνεπειών στο περιβάλλον και ήδη. Έχει ξεκινήσει την συνεργασία με τα με ηλία. Με του επίτροπου επίση. Όσον το χαρτοφυλάκιο έχει σχέση με τα θέματα αυτά την ανάπτυξη, για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και βέβαια συνεργασία με την Καθιάστον και βέβαια του χρόνου πρόκειται να κατεβάσουμε νομοθετική πρόταση η οποία θα βασίζεται σε αυτή την ανακοίνωση οπότε και εσείς θα έχετε καλυφθεί όσον αφορά το με πόσο σοβαρό τρόπο αντιμετωπίσαμε αυτό που μα αναθέσατε. Δηλαδή, μια ικανότητα αντίδρασης, σοβαρή αποτελεσματική από πλευράς Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ Επίτροπε Γεωργίευα για αυτό το σαφές μήνυμα προς την Επιτροπή σχετικά με το συντονισμό των ικανοτήτων και σχεδιασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαριθμίσατε τις καταστροφές που θρυνήσαμε το 2010 και τα μηνύματα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά για το μέλλον. Άρα χρειάζεται συντονισμός και η καλύτερη δυνατή αντίδραση. Σειρά συναδέλφων ζήτησαν το λόγο. Πρώτος ο Κρήτον Αρσένης. Παρακαλώ. Thank you very Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε. Σας καλωσορίζω στην Επιτροπή μας και σας συγχαίρω για την υπευθυνότητα που δείχνετε στην ε, διεκπαιρέωση των καθηκόντων σας και στο Πακιστάν, όπως ε, φάνηκε. Για να μην πω ιδιαίτερα στο Πακιστάν, που ήταν ιδιαίτερα σοβαρή η κατάσταση και σας συγχαίρω για τις ιδέες που παρουσιάσατε για την επερχόμενη ανακοίνωση. Συμφωνώ ότι οι ιδέες αυτές κινούνται προς σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να εστιάσω μόνο σε κάτι που δεν μου είναι σαφές. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα πρόληψης των ανθρωπιστικών κρίσεων. Ξέρουμε ποιες είναι οι πιο ευάλωτες χώρες. Και υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι ευάλωτες λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ξέρουμε ότι υπάρχουν χώρες που θα πληγούν τα επόμενα χρόνια δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί τους. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι και ευθύνη της Επιτρόπου Χάντεγκαρτ και άλλων επιτρόπων, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα των ανθρωπιστικών κρίσεων. Ε, υπάρχει κάπου η, η έννοια της πρόληψης των ανθρωπιστικών κρίσεων. Γιατί έχουμε διάφορα σενάρια για τις επόμενες κρίσεις. Επίσης σας συγχαίρω για την ιδέα σα να χρησιμοποιήσετε την αναδάσωση ω εργαλείο, ούτω ώστε να μην ξανά συμβούν αυτέ οι πλημμύρε όπω αυτέ στο Πακιστάν, Φερρυπίν. Θα πρέπει το οικοσύστημα να γίνει πιο ανθεκτικό. Θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό. Θα πρέπει να βοηθήσουμε, να το προστατεύσουμε, ούτω ώστε να ενδυναμωθεί για να αποφευχθούν διάφορε θεομηνίε και καταστροφέ Και να διδαχθούμε από τις κρίσεις, ούτως ώστε να μην επαναληφθούν. Έντιτα Στρέλα. Ευχαριστώ την Σέμι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Κύριε Επίτροπε, σας συγχαίρω και εγώ για την πολύ σαφή και πλήρη παρουσίαση που μας κάνατε. Για αυτή την πολύ ρεαλιστική διάγνωση της κατάστασης στην Ευρώπη αλλά και στο εξωτερικό. Συμφωνώ και με την άποψή σας ότι οι καταστροφές επαναλαμβάνονται όλο και πιο συχνά και είναι όλο και πιο δυνατές αυτές οι θεομηνίες. Οι ειδικοί που ασχολούνται με τις κλιματικές αλλαγές προβλέπουν ότι στο μέλλον τα πράγματα θα επιδεινωθούν. Με αυτό το δεδομένο, εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια πρόληψη, να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή, αλλά και να δράσουμε όταν και όπου παρουσιάζονται αυτές οι θεομηνίες. Θα πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό έγκαιρης παρέμβασης, έγκαιρης αντιμετώπισης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά είναι σημαντικό και για τη βοήθεια που χορηγούμε σε τρίτες χώρες. Κυρία Επίτροπε, μιλήσατε για την έκθεση Φερέιρα που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Στην έκθεση αυτή Κάνουμε προτάσεις που είχαν ήδη εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και στη δική μου έκθεση, στην έκθεση που είχα ετοιμάσει εγώ. Εγκρίσαμε, εγκρίναμε λοιπόν την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την ξηρασία και την απερίμωση και επίσης ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια οδηγία για την πρόληψη και τη διαχείριση των πυρκαγιών. Αυτό είχε εγκριθεί το 2006. Τώρα, υιοθετήσαμε και εντάξαμε αυτές τις προτάσεις στην έκθεση της περασμένης εβδομάδας. Θα ήθελα να μου πείτε, εσείς από πλευρά σας, τι κάνατε, τι προθέσεις έχετε σε σχέση με αυτές τις προτάσεις που παρουσίασε και ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Edith. Κάρμεν Γιάν Πράμβιν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο για τη συμβολή της στην απόψινή συζήτηση. Όπως και οι άλλοι συνάδελφοι, θέλω και εγώ να τονίσω την σημασία της πρόληψης, ιδιαίτερα για τα δάση. Πολλές καταστροφές οφείλονται σε βιολογικά αίτια. Συγκεκριμένη ερώτηση τώρα, που αναφέρεται σε κάτι που θεωρώ ότι είναι και δική σας αρμοδιότητα και αρμοδιότητα του συναδέλφου Πίμπαλκ. Στην Τανζανία υπάρχουν ε, σχέδια σε σχέση με τη χλωρίδα και πανίδα εκεί. Προτίθεται η Κομισιόν να παρέμβει και να προσφέρει εναλλακτικές οι οποίες θα πρέπει να είναι σε πολιτικό επίπεδο, ούτω ώστε να αποφευχθούν να χτίσουν δρόμους σε περιοχές, για παράδειγμα, που δεν επιτρέπεται ή είναι προτιμητέο να γίνουν αλλού. Υπάρχουν και, έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις να κάνω και θα ακολουθήσουν και άλλοι συνάδελφοι. Είστε υπεύθυνοι για την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση των κρίσεων. Αυτά είναι οι δύο όψεις του νομίσματος όταν έχουμε μια καταστροφή. Επιτροπή Ανάπτυξης και Επιτροπή ε, Περιβάλλοντος για τα ανθρωπιστικά και την αντιμετώπιση κρίσεων. Ε, έχουμε δύο ε, οργανισμούς, έχουμε μία για την αντιμετώπιση, πώς δομούνται όλα αυτά. Επίσης, Είπατε ότι έχετε εφεδρίες εις ό,τι αφορά την ικανότητα που υπάρχει για αντίδραση σε τέτοιου είδους φαινόμενα σε περιφερειακό, τοπικό επίπεδο κλπ. Πώς θα χρηματοδοτηθεί αν υπάρχει ας πούμε πολιτική προστασία ή πυροσβεστική σε μια περιοχή και έχει εφεδρίες μπορεί να υπάρξουν προβλήματα ε, διαχείρισης γιατί εδώ υπάρχουν δαπάνες ε, συγκεκριμένα κότι θα είναι, θα, κόστη, θα είναι κοινοτική χρηματοδότηση, θα αναλάβει ο καθένας σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, ε, αν δούμε τη συνθήκη της Λισαβόνας που έπρεπε να την ξέρω πολύ καλά, στο άρθρο 214 λέει, μιλάει για ε, μια ειρηνευτική δύναμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, υπάρχει σκέψη να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, αυτά από μένα καταρχήν και μπορείτε να απαντήσετε και μετά θα ρωτήσουν και άλλοι συνάδελφοι. Ναι, ε, ε, θα, θα, απαντήσουμε, θα απαντήσετε πρώτα σε αυτό το γύρο ερωτήσεων και μετά θα ακολουθήσουν και άλλες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ καλές παρατηρήσεις και ερωτήσεις σας. Καταρχήν το θέμα της πρόληψης. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε την αύξηση της συχνότητας και της έντασης των καταστροφών χωρίς μεγάλη εστίαση στην ετοιμότητα και την πρόληψη. Οπωσδήποτε έχουμε πολλά στοιχεία, τεκμηριωμένα στοιχεία και αποδείξεις ότι η επένδυση στην ετοιμότητα και την πρόληψη ε, ε, αποδίδει πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάμε για αντίδραση σε ε, καταστροφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο μιλάμε για ετοιμότητα, πρόληψη από αντίδραση και αποκατάσταση και ανάδραση, feedback, ούτως ώστε να βελτιώσουμε την επόμενη φορά τις αντιδράσεις μας και το τι θα κάνουμε γενικά. Το Πακιστάν ήταν μια ξεκάθαρη περίπτωση, γιατί το Πακιστάν είναι από τις 30 ε, πιο ευάλωτες χώρες εις ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματος. Δηλαδή, όλα τα έχει. Ε, επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή, έχει μεγάλη δημογραφική ανάπτυξη, μεγάλη αστιφιλία και ρήμωση της υπαίθρου, όταν ε, πήγα στο Πακιστάν είδα κατεστραμμένα χωριά από τις πλημμύρες σε περιοχές όπου δεν θα έπρεπε να έχουν κτίσει, να, υπάρχει, ε, να υπάρχει δόμηση. Καταστρέφει λοιπόν η πλημμύρα τη, τα σπίτια και αν δεν αλλάξει η συμπεριφορά τους ε, θα ξανακαταστραφούν. Επίσης η απερίμωση των δασών παίζει ρόλο και στο Πακιστάν και αλλού. Η IT, στην IT η απερίμωση, των, η αποψήλωση των δασών δημιουργεί κατολισθήσεις, δεν συγκρατούνται τα εδάφη. Αν είχε τα δάση της, αν είχε τη χλωρίδα που είχε παλιά η IT, θα, είχε, θα είχαν αποφευχθεί τα χειρότερα. Η δουλειά πάνω λοιπόν στην πρόληψη, πάνω στην ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων, είναι επιτακτική. Αρχίσαμε ήδη να κάνουμε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι πολύ γνωστό ότι ήδη σήμερα από τον προϋπολογισμό για την ανθρωπιστική βοήθεια δαπανούμε 6 με 8% έτσι δεν είναι, έτσι δεν τα υπολογίσαμε Πίτερ την τελευταία φορά για την ετοιμότητα. Το 6 με 8% του προϋπολογισμού για την ετοιμότητα χρηματοδοτήσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι για την ε, ετοιμότητα κατά των καταστροφών σε χώρες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε φυσικές καταστροφές. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ε, μειώσουμε τις ανθρωπιστικές καταστροφές, ενισχύοντας την ικανότητα της κοινωνίας να ε, αντιδρά. Και συνεργαζόμεθα με τον Επίτροπο Υπεύθυνο για την Ανάπτυξη και την Κόνι Χέντεγκαρτ για την υπεύθυνη Επίτροπο για την Κλιματική Αλλαγή για να δούμε πώς μπορούμε να ε, συμβάλλουμε όλοι και από όλες τις πλευρές στην ανθεκτικότητα, δημιουργία αντοχής στις κλιματικές αλλαγές. Γιατί είναι πολύ επίπεδο το καθήκον και μόνο μαζί μπορούμε να δουλέψουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και η Ευρώπη μαζί με άλλες χώρες και περιοχές του κόσμου για να κάνουμε τη διαφορά. Για την ανακοίνωση τώρα αυτή θα επικεντρωθεί στην απόκριση στις καταστροφές από άποψη διαχείρισης πόρων αλλά θα ενταχθεί σε αυτή τη συνολική προσέγγιση και έτσι θα την δείτε, με την έννοια δηλαδή ε, πρόληψη, ετοιμότητα, απόκριση, αποκατάσταση, feedback, ανάδραση. Ε, κάνατε και μια ερώτηση για την οδηγία για τα δάση. Αυτή είναι μια ερώτηση που μου την έκαναν και στην ακρόαση επίσης. Η προσέγγιση μας τώρα, και αφότου ήρθα εδώ έμαθα περισσότερα για την προσέγγιση μας, ε, εμείς ε, έχουμε μια προσέγγιση πολλαπλών κινδύνων. Τι σημαίνει αυτό. Ετοιμάζουμε κατευθυντήριες γραμμές για ε, μελέτη επίπτωσης κινδύνων για κάθε κατηγορία κινδύνων ή επικινδυνότητας, αν θέλετε, συμπεριλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών που θα συμπεριληφθούν ως προτεραιότητα στο πρόγραμμα ορθών πρακτικών για την αντιμετώπιση των καταστροφών που κάνουμε τώρα και σε ό,τι αφορά την ανάγκη για πρόσθετη νομοθεσία, το Μάρτιο του 2010 η Κομισιόν άρχισε μια συζήτηση για το μέλλον μιας ε, δράσης κοινοτική για την προστασία των δασών και για την ενημέρωση στον τομέα. Υπάρχει διαδικασία διαβούλευσης που έκλεισε τον Ιούλιο του 2010 ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι δηλαδή η διαβούλευση. Τώρα γίνεται μια αξιολόγηση του τι προέκυψε από αυτές τις διαβουλεύσεις και πάνω σε αυτή τη βάση στις αρχές του 2011 συγγνώμη, θα ε, υποβληθεί η πολιτική πρόταση. Και οι φωτιές στα δάση είναι ένα θέμα μεταξύ πολλών. Θα γίνει λοιπόν αξιολόγηση κινδύνου για τις δασικές πυρκαγιές καθοδήγηση αντολισμός για ορθές πρακτικές, ιδιαίτερα στην καταπολέμηση και πρόληψη δασικών πυρκαγιών και θα δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος και τι, τι νομοθετικό κενό πρέπει να κλείσουμε. Αυτά θα γίνουν αρχές του 2011, αλλά η προπαρασκευαστική εργασία και οι διαβουλεύσεις έχουν ολοκληρωθεί. Ε, επίσης, Τώρα για την Τανζανία, ε, για το, τη χάραξη δρόμου εκεί. Αν πρόκειται για κατασκευή οδού στην καρδιά πολύτιμου δάσους, μπορεί η καταστροφή να είναι μεγαλύτερη από τα ωφέλη που θα δώσει το έργο αυτό της οδοποιίας. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά το έχουμε ξαναδεί αυτό. Ε, κατασκευή δρόμου, οικονομικές δραστηριότητες εκεί και πολλές φορές ε, είναι οι επιπτώσεις χειρότερες από ό,τι αρχικά είχαν υπολογιστεί. Θα το ερευνήσω το θέμα και θα επανέλθω την επόμενη εβδομάδα να σας απαντήσω. Τώρα, ανθρωπιστική βοήθεια, πολιτική προστασία. Πώς θα συγκεράσουμε τα δύο. Είναι μία από τις περιπτώσεις αυτές ε, όπου ο γαμπρός νύφη δεν ήθελαν το γάμο, εξαναγκάστηκαν να παντρευτούν όμως. Δηλαδή είναι γάμος από συνοικέσιο ας το πούμε. Όταν όμως έγινε ο γάμος, αφού παντρεύτηκαν, τα, πήγαν πολύ καλά και ευτύχησε η οικογένεια. Και πραγματικά μου κάνει ε, ε, κατάπληξη πόσο καλά προχωρεί το πρόγραμμα αυτό. Εγώ περίμενα ε, περισσότερα θεσμικά προβλήματα και αντιδράσεις, αντιστάσεις. Αλλά η πραγματικότητα φέτος έδειξε άλλα. Ήταν πραγματικά ένα τεράστιο καθήκον αυτό που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, να βοηθήσουμε τον κόσμο ε, που είχε ανάγκη. Οι δύο ομάδες λοιπόν ανθρωπιστικής βοήθειας από τη μια και πολιτικής προστασίας από την άλλη συνεργάστηκαν αποτελεσματικότατα επί τόπου. Και μετά βέβαια οι επιπτώσεις άρχισαν να ε, σημειώνονται και προς τα πάνω και προς τα κάτω γιατί και αυτό εδραίωσε την ε, ε, ολοκληρωμένη δράση. Στο Πακιστάν υπάρχει τώρα μια ομάδα. Ε, η βοήθεια δηλαδή συντονίζεται και για την ανθρωπιστική και για την πολιτική προστασία. Ως εδώ καλά θέλουμε να φροντίσουμε και να εξασφαλίσουμε ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί και αυτό στηρίζεται από την ανακοίνωσή μας. Για το άρθρο 2.14 είπατε μου φαίνεται για την, ε, το σώμα αυτό των εθελοντών. Αρχίσαμε τις προπαρασκευαστικές εργασίες και αυτή τη βδομάδα, μου φαίνεται την πέμπτη αυτή τη βδομάδα, θα αρχίσει και επίσημα η διαδικασία αυτή για να δούμε πώς θα συσταθεί το σώμα αυτό. Δεν θέλουμε να χάσουμε τον επόμενο χρόνο που είναι ε, το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντών, αλλά ούτε θέλουμε ε, μεσοβέζικες λύσεις. Ε, θα περάσω μίσος από πιλωτική φάση. Το 2011 θα είναι σε πιλωτική φάση και μικρότερη κλίμακα και μετά θα το αναπτύξουμε τις επόμενες χρονιές για να έχουμε προστιθέμενη αξία ε, από την κοινότητα των εθελοντών και βέβαια να ε, προαχθούν και οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μου φαίνεται απάντησα στις ερωτήσεις αυτού του γύρου. Α, και το τελευταίο, ποιος θα, θα πληρώσει τις ικανότητες που είναι σε εφεδρεία. Α, ε, ζητώ συγγνώμη, το ξέχασα. Ερώτησε για ένα εκατομμύριο ευρώ, 60.000 ευρώ μάλλον. Θα, μπορέ, θα προσπαθήσω να σας απαντήσω όσο πιο ακριβώς μπορώ αυτή τη στιγμή. Αυτό που προτείνουμε είναι τα κράτη-μέλη να διαθέσουν κάποια μέσα εθελοντικά για να χρησιμοποιούνται σε κοινοτικό επίπεδο. Τα κράτη-μέλη πληρώνουν για αυτά τα μέσα, για αυτές τις εφεδρίες. Και το όφελο για αυτού ποια είναι, η αμοιβαιότητα. Αν χρειαστούν δηλαδή αυτά τα μέσα, θα του βοηθήσουν άλλοι. Ήρθα σε επαφή με διάφορα κράτη-μέλη, ήρθα σε επαφή με του υπεύθυνου για τα συστήματα πολιτική προστασία και μέχρι στιγμής υπάρχει ενθουσιασμό σε πολλά κράτη-μέλη για να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια υπάρχουν και κάποια άλλα που έχουν διαφορετικές απόψεις. Υπάρχουν δύο στοιχεία πάντως που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Το ένα είναι οι μεταφορές. Αν οι χώρες συγκεράσουν τα μέσα τους για να μεταφερθούν κάπου αλλού, τότε περιμένουν ότι κάποιος θα βοηθήσει την προσπάθειά τους. Δεύτερον, αν διαθέσουμε κάποια κοινωτικά μέσα για να καλύψουμε κάποιες τρύπε, φυσικά αυτά κοστίζουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δημοσιονομικά είμαι πολύ συντηρητική. Πιστεύω ότι οι φορολογούμενοι μας περιμένουν να ξοδέψουμε μεγάλη σύνεση και τσιγκουνιά, αν θέλετε, κάθε ευρώ. Και οτιδήποτε ξοδέψουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει πραγματικά να αξίζει. Αλλά δεν θέλω να σας πω ότι δεδομένου το προβλήματος μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο. Υπάρχει κάποιο κόστος και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να το καλύψουμε αυτό το κόστος, αυτή η δαπάνη. Ούτως ώστε να συγκεραστούν όλες αυτές οι εθνικές προσπάθειες και τα εθνικά μέσα και να δημιουργήσουν μία κοινοτική απόκριση. Καταρχήν πρέπει να κάνουμε κάποιες προτάσεις πολιτικής και αν υπάρξει υποστήριξη θα κάνουμε μία πλήρη αξιολόγηση για το κόστος. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, να καλωρίσω τον κύριο Πέτερ Τσάνι, ο οποίος είναι ο διευθυντής του ΕΚΟ και οι συνεργάτες του, ε, Έχουμε και εδώ δύο θέσεις, αλλά και εκεί καλά είστε. ακούμε με χαρά ότι τρέχει καλά το πρόγραμμα. Ε, δηλαδή αυτή, αυτός ο συγκερασμός των αρμοδιοτήτων σε μία αρχή πάει καλά. Προφανώς τριβές και δυσκολίες θα υπάρχουν, αλλά γενικά πάει καλά. Άλλες ερωτήσεις, πασάικο του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε που ήρθατε που ήσασταν τόσο λακωνικοί και που μιλήσατε για τα θέματα του χαρτοφυλακίου σας, που είναι αρκετά ευρύ, αλλά τα παρουσιάσατε με τρόπο πολύ συνοπτικό και σαφή. Μία συγκεκριμένη ερώτηση για τον κόλπο του Μεξικού. Και μια και αντιμετώπιση των κρίσεων είναι και δική σας αρμοδιότητα, το ερώτημά μου αφορά την αντιμετώπιση των κρίσεων μέσα στα ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα. Αυτό που συνέβη στο Μεξικό μπορεί να συμβεί και στα δικά μας ύδατα. Στο ψήφισμα που υιοθετήσαμε ζητάμε μια συνολική μονάδα που να αντιμετωπίζει όλα αυτά τα θέματα. Ε, σε ποιο βαθμό προωθείτε κάτι τέτοιο σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, προφανώς, αλλά εσείς πόσο το προωθείτε. Νομίζω ότι έχει γίνει ανάλυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχετε καταλήξει ότι έχουμε επαρκές δυναμικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η περιβαλλοντική πολιτική έκανε μεγάλο βήμα μπροστά με την πολλαπλή συμμόρφωση, το cross compliance ε, και τις ρυθμίσεις για τον, στο γεωργικό τομέα. Μπορεί να υπάρξει τώρα μια νέα προοπτική ανάπτυξης της ανθεκτικότητας ε, στην περιφερειακή πολιτική κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε να υπάρξει ανθεκτικότητα και απέναντι στις ε, φυσικές καταστροφές. Ε, συνήθως πλημμύρες είναι τα προβλήματα αυτά και υπάρχει και η οδηγία με την οποία, για τις πλημμύρες με την οποία κάναμε το πρώτο βήμα, αλλά ακόμα δεν είναι αρκετά ικανοποιητικό το νομοθετικό πλαίσιο, ούτως ώστε να επιτρέπει καλή αντίδραση στις καταστροφές. Στις κομισιόν εσείς θα καταβάλλετε προσπάθειες, ούτως ώστε να έχουμε πολλαπλή συμμόρφωση για αυτές τις αντιδράσεις και προετοιμασίες που θα χρηματοδοτούνται από κονδύλια της Ένωσης και ε, μετά ε, και κονδύλια από τις περιφέρειες αλλά και από τον γεωργικό τομέα. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν μια ε, ανθεκτική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θα είναι καλός ο λόγος να πάνε των κονδυλίων αυτών. Επίσης, υπήρξε η ιδέα για κάποια προστασία ασφαλιστική σε περίπτωση πλημμυρών γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχει ασφάλεια για τέτοιας μεγάλης κλίμακας καταστροφές. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο από την Κομισιόν το οποίο θα ασχολείται ακριβώς με αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Το, αυτό το τελευταίο αναφέρεται και στο ψήφισμά μας του Σεπτεμβρίου και θα αναφέρεται και στο επόμενο ψήφισμά μας δηλαδή ε, πώς μπορεί κανείς να καλύψει τις ζημίες, απώλειες. Πολλές φορές ε, η ασφάλεια είναι ελάχιστη ή ανύπαρκτη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια θα ενταχθεί στο δικό σας το χαρτοφυλάκιο. Τι ασφαλιστικές λύσεις μπορεί να ε, υπάρξουν τόσο ώστε να μην πληρώνει πάντα ο φορολογούμενος, αλλά να υπάρχουν συλλογικά συστήματα ε, που θα αναλαμβάνουν τον ασφαλιστικό κίνδυνο. Η Επίτροπος. Για το θέμα του κόλπου του Μεξικού. Από την αρχή δράσαμε σωστά. Όλοι οι επίτροποι που έχουν ευθύνη που συνδέεται με το πρόβλημα στο κόλπο του Μεξικού, ο, η Επίτροπος για το Περιβάλλον δηλαδή, και με επικεφαλή στον Επίτροπο Ότιγκερ, αλλά και η Επίτροπος Αλίας και εγώ ήρθαμε σε επαφή, συζητήσαμε. Κάναμε ειλικρινείς συζητήσεις και με τον ιδιωτικό τομέα. Μιλήσαμε έξω από τα δόντια για το πρόβλημα, για τις προσδοκίες μας, ο Επίτροπος Ότιγκερ με απόψεις που, στις οποίες συνεισφέραμε και εμείς θα ετοιμάσει μία ανακοίνωση για να δούμε πώς μπορούμε πραγματικά να ενδυναμώσουμε την περιβαλλοντική νομοθεσία στον τομέα αυτό, τόσο ώστε στα ύδατά μας να μην δημιουργηθούν τέτοια προβλήματα πετρελοκυλίδας και αν και οι νομοθετικές προτάσεις θα επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογή των σημερινών προτάσεων, είτε θα υπάρξουν νέε νομοθετικέ προτάσει. Θα δούμε, θα βολιδοσκοπήσουμε του ενδιαφερόμενου και θα δούμε τι αξίζει να προχωρήσουμε. Από αυτά που ακούσαμε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τον ιδιωτικό τομέα, δεν διστάζουμε και να ζητήσουμε πολλά και να είμαστε πολύ απαιτητικοί σε επίπεδο νομοθεσία. Γιατί αυτό που συνέβη στον κόλπο του Μεξικού θα μπορούσε να έχει συμβεί και στην Ευρώπη. Ευτυχώ δεν συνέβη βέβαια. Αλλά με ποιο τρόπο εμεί ετοιμαζόμαστε ούτω ώστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό είναι και θέμα πολιτική και τεχνολογική αξιολόγηση και τι σχετικέ προτάσει θα τι παρουσιάσουμε πολύ σύντομα. Θα τι δείτε κι εσείς. Υπάρχει και εδώ κάποιος από το γραφείο μου που ασχολείται με αυτό το θέμα. Στην αρχή δεν ήμουν σίγουρη για το πώς θα προχωρήσουμε, για το αν ο ιδιωτικό τομέα θα ενδιαφερθεί. Και στις πρώτες επαφές έδειξαν κάποιους δισταγμούς, αλλά τελικά εμείς συνειδητοποίησαμε ότι με αυτούς ή χωρίς αυτούς θα υπάρξει ενδυνάμωση της νομοθεσίας και νομίζω ότι τελικά προέκυψε και διάθεση για συνεργασία. Φυσικά στον ιδιωτικό τομέα διαφορετικές εταιρε... διάφορες επιχειρήσεις ή εταιρείε έχουν διαφορετικές απόψεις. Κάποιες είναι πιο πρόθυμες να βοηθήσουν, κάποιες λιγότερο. Αλλά ενδυναμώνουμε, εντατικοποιούμε τις ε, προσπάθειές μας. Τώρα, για την οδηγία για τις πλημμύρες και τη χρηματοδότηση. απογοητεύτηκα λίγο που είδα ότι οι χώρες χρησιμοποιούν με ανεπαρκή τρόπο τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, που έχουν στη διάθεσή τους. Και ελπίζω ότι φέτος το καλοκαίρι κάποιοι άκουσαν τον κόδωνα κινδύνου. Και όλο το χρόνο. Έχουμε, ερχόμαστε σε επαφή με κράτη-μέλη που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, ούτω ώστε να τα βοηθήσουμε να χρησιμοποιήσουν όλους τους διαθέσιμους πόρους. Και τα κράτη-μέλη το αναγνωρίζουν. Αναγνωρίζουν την ανάγκη να τους χρησιμοποιήσουν καλύτερα. Τώρα η ανησυχία μου εμένα είναι η εξή. Η πιο μεγάλη ανησυχία. Η ικανότητα απορρόφηση κονδυλίων για φυσικές υποδομές, που είναι μεγαλύτερη από την ικανότητα απορρόφηση κονδυλίων για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Θα πρέπει αυτά τα δύο πράγματα να εξισορροπηθούν κάπως. Γιατί δεν αρκούν μόνο οι υποδομές. Μερικές φορές οι πολιτικές και οι αποφάσεις είναι πολύ πιο σημαντικές από τις ίδιες υποδομές. Τι γη, α πούμε, θα χρησιμοποιήσουμε για αστική ανάπτυξη, ποια γη προστατεύεται για γεωργική χρήση και ούτω καθεξής. Εμείς για να προλάβουμε τις καταστροφές θέλουμε να συζητήσουμε περισσότερο, να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να εστιάσουμε περισσότερο στο θεσμικό και πολιτικό στοιχείο και επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών. Τα λεφτά υπάρχουν. Και τα γεγονότα που συνέβησαν μας δικαιολογούν και δικαιολογούν τη συνέχιση αυτής της πολιτικής για τον σχεδιασμό και στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Ε, δεν νομίζω να παρεκκλίνουμε από αυτή την ρότα. Τώρα, για τις ασφάλειες. Και στην, ανθρωπιστική βοήθεια, εγώ μίλησα με τους συναδέλφους μου ε, για αυτό το θέμα και μου είπαν ότι δεν πιστεύω ότι είναι βιώσιμη λύση αυτή. Έχουμε 800 εκατομμύρια ευρώ μέχρι ένα δις. Σε περίπτωση που χρησιμο... φτάνουμε και στο ένα δις αν χρησιμοποιήσουμε και τα λεφτά του αποθεματικού. Αλλά φέτος, στα μέσα του Αυγούστου, ξεμείναμε από λεφτά. Γιατί υπήρχαν τόσες πολλές ανθρωπιστικές καταστροφές ανά τον κόσμο. Το να έχουμε τώρα μια, ένα οικονομικό σχεδιασμό που να μην βασίζεται στον προϋπολογισμό και στο αποθεματικό, θα πρέπει να έχουμε και ένα σχέδιο για τις ασφάλειες, ούτως ώστε τα χρήματα να επενδύονται που έχουμε, ούτως ώστε οι χώρες που αντιμετωπίσουν τις περισσότερες, τους περισσότερους κινδύνους για θεομηνίες και κάθε χρόνο μπορούμε να το προβλέψουμε, γιατί ας πούμε του χρόνου θα πρέπει να προβλέπουμε το Σουδάν ότι θα αντιμετωπίσει θεομηνίες. Να είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Απλώς δεν έχουμε αυτή την οτροπία να χρησιμοποιήσουμε ένα τμήμα του προϋπολογισμού μας, ούτως ώστε να απελευθερώσουμε άλλα κονδύλια και η δυνατότητα χρηματοδότησης που έχουμε να συνοδεύει τη δυνατότητα δαπανών που έχουμε. Νομίζω ότι αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε ε, για το πώς θα ξαναδούμε το θέμα του οικονομικού σχεδιασμού για τη χρηματοδότηση των θέματων αυτών. Πρέπει να συζητήσουμε για το πώς θα έχουμε ένα οικονομικό σχεδιασμό που εντάσσεται σε αυτό το σενάριο. Και βέβαια το βασικό που πρέπει να εξετάσουμε είναι το θέμα της έλλειψης πρόβλεψης για να είμαστε ευέλικτοι και έτοιμοι. Είναι πολύ σημαντικό να λειτουργούμε με σενάρια. Frau das war... Κυρία Επίτροπε Γεωργίευα, αυτή ήταν η αρχή της συνεργασίας μας ως Επιτροπή Ανάπτυξης, ε, περιβάλλοντος. Ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων που είχαμε. Ε, βεβαίως προσβλέπουμε στην ανακοίνωση τις, ε, τους επόμενους μήνες και βέβαια σε νομοθετικό επίπεδο είναι πολύ σημαντικά αυτά που θα περιμένουμε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι του χρόνου είναι το ε, έτος των ε, εθελοντών. Οπότε ένα τέτοιο σώμα εθελοντών θα ενδιαφέρει πολύ τους νέους. Θα έχει απήχηση σε ανθρώπους που θέλουν να ε, βοηθήσουν και να αφοσιωθούν σε ένα σκοπό. Ακούσαμε ότι η ευελιξία είναι σημαντική και πρέπει να υπάρχει και στον προϋπολογισμό. Ε, αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει και με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Προϋπολογισμών να το συζητήσουμε και να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να προβλέψουμε κάποια πράγματα και να είμαστε έτοιμοι να μην βρεθούμε μπροστά σε άδεια ταμεία όταν χρειαστεί βοήθεια. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτησή μας αυτή και οπωσδήποτε μετά την ανακοίνωση θα ειδωθούμε πάλι και μετά τις νομοθετικές σας προτάσεις. Ε, καλή επιτυχία μέχρι την επόμενη φορά. Ευχαριστώ. Ε, όποτε θέλετε θα με φωνάξετε και θα έρθω. Ωραία. Προχωρούμε στο σημείο 5 που είναι μια προφορική ερώτηση από τους συναδέλφους Κρήτων Αρσένη, Κορίν Λεπάζ, Λίντα Μακέιβεν, Σύρπα Πιέτη Κάινεν, Καρτί Καλιοτάρα, Ρόσμπαχ, σχετικά με την ε, ασφαλτούχο άμμο και τις αλλαγές στην χρήση της γης και την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων. Λοιπόν, κάποιος από τους επερωτώντες να μας κάνει την εισαγωγή. Ο Κρήτον Αρσένης, παρακαλώ. Thank you Mr. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ξέρουμε αυτό το θέμα πολύ καλά στην Επιτροπή. Το συζητήσαμε και τον Ιούνιο στην συνεδρίαση της Επιτροπής. Σήμερα, με βάση την τρέχουσα πρόταση της Επιτροπής, δεν υπάρχει αρχική τιμή για τις ε, εκπομπές στις ασφαλτούχες άμμους και ούτε και στους ε, ασφαλτούχους χιστόλυφους. Με το να μην έχουμε αρχική τιμή, θα χρησιμοποιούμε μια χαμηλότερη τελικά ε, τιμή, πολύ χαμηλότερη τιμή και επομένω θα επιδοτούμε αυτή τη δραστηριότητα. Η Κομισιόν μέχρι στιγμής είπε ότι καταργεί την τιμή που πρότεινε αρχικά, γιατί φοβάται ε, μήπως αμφισβητηθεί σε επίπεδο ΠΟΕ. Με βάση τους κανόνες όμως του ΠΟΕ, οι τιμές θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και στοιχεία. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Έχουμε τιμές για άλλα ορυκτά καύσιμα, που βασίζονται όμως σε μία απλή μελέτη. Από την άλλη, για τις ασφαλτούχες άμμος, ε, έχουμε 12 μελέτες που μιλούν για μία ε, μέση τιμή που είναι πολύ κοντά στην τιμή που πρότεινε η Κομισιόν. Επομένως, μπορούμε πολύ πιο άνετα να ορίσουμε μία αρχική τιμή για την ασφαλτούχο άμμο παρά για τα υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα. Παρότι εκεί πρότεινε η Επιτροπή. Παρότι οι τιμές που συζητούνται στις 12 μελέτες και που αρχικά προτάθηκαν από την Επιτροπή ε, είναι χαμηλές Μιλάμε για μια δραστηριότητα που θα καταστρέψει, καταστρέφει ήδη, αλλά και θα καταστρέψει και στο μέλλον, το 1 τέταρτο των άθικτων δασών αυτού του κόσμου. Μιλάμε για τα αρκτικά δάση του Καναδά, που είναι από τα πιο σημαντικά ε, και είναι δεξαμενή απορρόφησης διοξιδίου του άνθρακα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Η πρόταση τη Κομισιόν δεν μιλάει επίση για να συντελεστεί για τη χρήση τη γη. Δεν λαμβάνει υπόψη το κύκλο ζωή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στι μεταφορέ και δεν αξιολογεί τις εκπομπές, αυτές τις εκπομπές. Η πρόταση για να ξεπεράσουμε το επίπεδο του ΠΟΕ, ήδη είναι μια προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τα ορυκτά καύσιμα. Την τελευταία φορά εδώ στην Επιτροπή η Κομισιόν, μέσω του εκπροσώπου της, μας εξήγησε ότι τα κράτη-μέλη δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Να σας εξηγήσω αυτή την ιδέα η Κομισιόν βάζει ένα συντελεστή και ένα κράτος μέλος ή μάλλον μια εταιρεία η οποία παράγει ε, χρησιμοποιεί μάλλον τις ασφαλτούχες άμμους για την πετρέλαιο και έχει λιγότερες εκπομπές κατά την παραγωγή, μπορεί τότε να παρουσιάσει τα δεδομένα της και τότε θα αλλάξει ο συντελεστής για τη χρήση της ασφαλτούχου άμμου για την παραγωγή του πετρελαίου. Επομένως, υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής των συντελεστών όταν υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα. Και με αυτόν τον τρόπο επίσης μπορούμε να συλλέγουμε δεδομένα για να προχωρήσουμε πολύ πιο άνετοι στα επόμενα βήματα. Μετά από αυτά που μας είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, κάναμε μια συζήτηση, κοιτάξαμε τα έγγραφα των κρατών μελών και βρήκαμε ότι μόνο 10 κράτη-μέλη συμμετείχαν στη διαβούλευση. Πέντε από αυτά υποστήριζαν την υβριδική προσέγγιση και πέντε ήταν κατά της υβριδικής προσέγγισης. Αυτό το θέμα λοιπόν φαίνεται ότι δεν έχει συζητηθεί επαρκώς. Και τα κράτη-μέλη από ό,τι φαίνεται δεν θέλουν να το συζητήσουν. Καταλαβαίνουμε ότι μέχρι στιγμής η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποστηρίζει την υβριδική προσέγγιση. Αλλά εδώ ακούσαμε διαφορετικά πράγματα. Συγγνώμη, μάλλον η Γενική Διαθέση ε, Ενέργειας και η Γενική Διαθέση Περιβάλλοντος δεν συμφωνούν για την ε, υβριδική προσέγγιση. Επομένως, πέστε μας, ποια είναι η κατάσταση για την υβριδική προσέγγιση. Εάν δεν υπάρχει υποστήριξη για αυτή την προσέγγιση, γιατί από πλευράς Κομισιόν. Αυτό το επιχείρημα που λέει η Κομισιόν ε, για τον ΠΟΕ δεν ισχύει, διότι ο συντελεστής που έβαλε η Κομισιόν για τις ασφαλτούχες άμμους ε, υποστηρίζεται από, τις 12, από 12 ολόκληρες ε, μελέτες, ενώ οι άλλοι συντελεστές υποστηρίζονται από λιγότερες μελέτες. Επίσης, πέστε μου τι γίνεται με το συντελεστή για τη χρήση της γης στην οδηγία για τα καύσιμα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε τον Αρσένης για αυτή την εισαγωγή της ερώτησης στην Κομισιόν. Ζητήσαμε να έρθει από την Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και Κλίματος ο κύριος Σόουν και ο κύριος Ότσον ε, είναι οι εκπρόσωποι των δύο γενικών διευθύνσεων. Κύριε Όουεν, θέλετε να λάβετε εσείς πρώτος το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Αρσένη για την εισαγωγή με τόση ακρίβεια στο θέμα. Θα απαντήσω αντίστροφα. Θα μιλήσω πρώτα για τα υβριδικά και μετά για τις ασφαλτούχους άμμους. Ε, χαίρομαι που είχα τη δυνατότητα να έρθω και να μιλήσω για το συνεχιζόμενο έργο μας σε σχέση με την οδηγία για τα κάψιμα την αναθεώρηση. Για το 7α ακόμα δεν έχει υποβάλει πρόταση για την ποιότητα. Υπάρχουν ε, έγγραφα διαβούλευση, συνεχίζονται οι συζητήσεις με εμπλεκομένους και τα κράτη-μέλη. Περαιτέρω διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Μέχρι τώρα από τα έγγραφα φαίνεται ότι οι υπηρεσίε τη Κομισιόν εξέτασαν την υβριδική προσέγγιση λεπτομερώ. Αυτά είναι στοιχεία από το έγγραφο με του εμπλεκόμενου που δημοσιεύτηκε το 2009 Διάφορε εναλλακτικέ τον Ιανουάριο του 2010 παρουσιάστηκαν και υπάρχει και το έγγραφο των επιλογών των εναλλακτικών που παρουσιάστηκε στα κράτη-μέλη το Μάρτιο του 2010. Συνεχίζεται η διαδικασία όπως σας είπα, εξετάζεται το θέμα. Όποια και αν είναι η τελική θέση είναι σημαντικό η προσέγγιση μας στα εφαρμοστικά μέτρα να είναι ισορροπημένη και επαρκή. Αυτό αναγνωρίστηκε από του συνομοθέτε που επέλεξαν να μην επαναλάβουν την ε, ε, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό για τα ορυκτά καύσιμα. Θέλουν η μεθοδολογία να αναπτυχθεί συγκεκριμένα ε, ε, για τα καύσιμα εγκεκριμένη από την Επιτροπολογία. Οποιαδήποτε προσπάθεια που θέλει να συμπεριλάβει τη φάση της εξόρισης, διήλυσης, θέτει δύσκολα θέματα υπολογισμού. Πρέπει να θυμόμαστε ότι τα ε, βήματα αυτά στον κύκλο ζωής ε, δημιουργούν 15% μόνο των ε, εκπομπών. Πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις εκπομπές ασφαλτού χωνάμων. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε μια μέθοδο η οποία θα οδηγήσει σε σωστή και ικανοποιητική μείωση των εκπομπών του πράσινου άνθρακα. Το εξετάζουμε αυτό. ισότι ό,τι αφορά τι νομοδοτήσει των κρατών μελών, η δημόσια διαβούλευση πάνω σε αυτό το θέμα ε, έδωσε απαντήσει από 13 κράτη-μέλη. Δύο ερωτήματα ετέθησαν σε σχέση με την προτιμόμενη μέθοδο υπολογισμού του πράσινου άνθρακα. Έξι θέλουν τη μέθοδο σημαντική τιμή, οι άλλοι ε, δύο θέλουν την υβριδική. Επίσης, ε, θα πρέπει να ε, υπάρχει ε, μια οδηγία η οποία θα συμπεριλαμβάνει και την μέθοδο για τα ορυκτά καύσιμα. Δύο κράτη-μέλη υπέρ, έξι κατά. Το Μάρτιο του 2010 παρουσιάστηκε το κείμενο των εναλλακτικών με οκτώ εναλλακτικέ μόνο συμβατικής τιμής ή και υβριδικής. Τα πρακτικά έδειξαν ότι 10 κράτη-μέλη θέλουν μια συμβατική τιμή μαζί με μια ρήτρα επανεξέτασης. Μετά, τρία κράτη-μέλη υποστήριξαν τις συμβατικές τιμές. Ένα μόνο κράτος-μέλος διαφώνησε ε, ξεκάθαρα με την προσέγγιση αυτή. Εις ό,τι αφορά τώρα τις ασφαλτούχους άμμους, η Κομισιόν δεν έχει κάνει διεξοδική αξιολόγηση σε σχέση με τις ε, άμμους αυτές και τα κάψιμα. Αυτή η μέθοδος ε, θα εξετάστηκε σε σχέση, ε, από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Τώρα το κονσόρτσιουμ που αρμόδιο κονσόρτσιουμ ε, ε, ετοιμάζει μια έκθεση. Υπάρχουν πολλές εκθέσεις επίσης που δίνουν πρόσθετες πληροφορίες για τις ασφαλτούχους άμμους. Η Κομισιόν τώρα σχεδιάζει τα εφαρμοστικά μέτρα. Όμως σε μια, ε, τον περασμένο Ιούλιο απίφθινε στις 14 Ιουλίου μια επιστολή προς τα κράτη-μέλη ούτως ώστε να ε, προχωρήσουν στη συμβατική τιμή ε, φόσον θα έβρισκε σύμφωνα τα κράτη-μέλη το ταχύτερο δυνατόν. Μετά θα ακολουθούσαν τα εφαρμοστικά μέτρα προς τα κράτη-μέλη. Μέχρι πριν από το τέλος του 2011 η Κομισιόν θέλει να ολοκληρώσει το θέμα όταν θα έχουμε και αποτελέσματα από τις μελέτες ε, που έχουν ανατεθεί. Τέλος, ε, ε, για την αλλαγή χρήσης γης. Ε, και αυτό θα πρέπει να το δούμε, μας έχει ε, απασχολήσει και εμάς και άλλους. Σε σχέση με το ζήτημα αυτό, ασφαλτούχους άμμους και εκπομπές από αλλαγή χρήσης γης, ε, η περιβαλλοντική υπηρεσία θεωρεί ότι η, ε, στην εξόριξη, στον Καναδά για παράδειγμα, μπορεί 0,6 γραμμάρια ε, ανά μεγατζάουλ διοξιδίου του άνθρακα να είναι το αποτέλεσμα. Αυτό είναι λιγότερο από το 1% του, των εκπομπών από, για, για πετρέλαιο ή, βενζι, ή δίζελ. Ε, έτσι λοιπόν ε, στις υπόλοιπες περιπτώσεις η εξόρυξη in situ είναι η μεγαλύτερη ε, πηγή εξόρυξης ασφαλτούχων άμμων στον Καναδά. συνολικά εξετάσαμε την υβριδική μέθοδο, δεν έχουμε καταλήξει ακόμη και οι ασφαλτούχοι άμοι έχουν ε, ληφθεί επαρκώς υπόψη στις μελέτες μας που συνεχίζονται και στις διαβουλεύσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει να παρέμβει ο κύριος Χάτσον. Αν όχι, ο Πατ Άικοντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Όγον για τόσο μας εξήγησε, για τόσο μας απαντήσατε. Σε συνέχεια τον όσων ακούσαμε, το πιο σημαντικό είναι το timing, ο χρονισμός και θα πρέπει η Επίτροπος επίσης να τηρήσει την υπόσχεσή της, τη δέσμευσή της και να δούμε τι θα γίνει, γιατί ε, μέχρι τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η Επιτροπή, περιμένοντας και τις ε, σχετικές μελέτες. Θα πρέπει όμως να μην ξεχνούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα προς τους επενδυτές. Αυτό γίνεται τώρα. Μήπως ξέρετε, στο, έχουμε 379 δις ευρώ που θα επενδυθούν σε ασφαλτούχο άμμο. 3,79 δις θα επενδυθούν σε ασφαλτούχο άμμο και εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στείλει τώρα το σωστό μήνυμα ότι δηλαδή πρόκειται να ορίσουμε μία τιμή, τότε θα προχωρήσουν οι επενδυτές. Και προχωρήσουμε εν ώψη του 2011 σαν ορίζοντα, θεωρώντας ότι θα, γίνει, γίνουν σχετικές απαγορεύσεις κλπ. Άρα, δεν μιλούμε εδώ για κάποιο είδους δημόσιο έγγραφο, μιλούμε για κάποιες επιστημονικές εκθέσεις. Άρα θα πρέπει όλα αυτά να κατατείνουν στον ίδιο στόχο. Στο κατά πόσον δηλαδή μολύνει όχι η συγκεκριμένη άμμος, η ασφαλτούχος άμμος. Και επομένως να ξέρουν οι επενδυτές κατά πόσον είναι σωστό ή όχι το να επενδύουν σε αυτό το υλικό. Κρήτονα. Πάρα πολύ χαίρομαι που βλέπω ότι κάπω άλλαξε ρότα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλαξε γνώμη και καταλαβαίνει τώρα ότι η βρυδική προσέγγιση θα προληφθεί περισσότερο απόψη που παλιότερα ήταν αυτό το οποίο είχε απορριφθεί από τα κράτη-μέλη και ότι τώρα κινούμεθα ε, προ καθεσμό κάποια οριακή τιμή για την ασφαλτούχο άμμο. Τώρα το χρονοδιάγραμμα. Μιλούμε για τέλη του 2011, οπότε τότε ίσως δεν είναι το σωστό το μήνυμα που θα να δώσουμε προς τους επενδυτέ Ίσως να επιδοτηθεί κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα και να κινούμε προς τη λύση της Μαδαγασκάρης. Δεν ξέρω πόσο σίγουρη είναι από Καναδά, Μαδαγασκάρ και λοιπόν που να δούμε επομένω τώρα. Τι θα γίνει με την εξασφάλιση των επενδύσεων σε σχέση με την πρώτη ύλη που θέλουμε να, να, να πάρουμε ε, γιατί είπαμε ότι τελικά δεν έχουμε την πολυτέλεια και το περιθώριο του να στείλουμε το λάθος μήνυμα. Επομένως να οριστεί το ίσως κύριε οριακή τιμή. Well, uh, I think, Owen, if you want to have a floor for a reply, that's okay. Commission. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ 100% ότι η βιομηχανία θέλει έναν ε, ορατό ορίζοντα να προγραμματιστεί και άρα θα βρούμε όσο γίνεται πιο συγκεκριμένοι για το τι θα πρέπει να κάνουν στο μέλλον εκείνοι. Και ξέρω ότι έχετε και αύριο σε σχέση με τις φοβές διοξιδίου και τα, και τα οχήματα για εμπορικούς, εμπορικές κάποια ψηφοφορία. Δεν είναι και τόσο μακριά ο του 2011, οπότε θα πρέπει όντω να έχει τεθεί για την ασφαλτούχα μου κάποιο, κάποιο τιμή και αυτό θα είναι μήνυμα προ την βιομηχανία και σήμερα του λέμε ότι δεν έχουμε ε, κάποια τιμή να σα δώσουμε, ε, όμως αυτό ε, το, το, το, το, μελετούμε σε σχέση και ε, με τις μελέτες που γίνονται, ούτως ώστε να μπορούμε να προγραμματίσουμε τις ε, επενδύσεις και τελικά θα υπάρξει ο ορισμός της τιμής και νομίζω αυτή είναι η απάντηση σε αυτό που ρωτήθηκε. Εδώ λίγη συζήτηση για αυτό το σημείο είναι ο κύριο Λίτερ. Το επόμενο θέμα. Ε, προέρχεται από τους βουλευτές Σάτου Χάσε και Κρίς Ντέιβις και αφορά τα όρια εκπομπών και μείωση σε θείο των καυσίμων πλοίων. Όμως οι συνάδελφοι δεν είναι εδώ. Υπάρχει κάποιος που τους αντικαθιστά. Α, ναι, υποσχέθηκαν ότι αντικαταστήσω, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Άρα καλύτερα να μην πω τίποτα και μετά στις δευτερολογίες να πω. πάντω. ζητούν συγγνώμη που δεν είναι εδώ οι συνάδελφοι. Ε, τα ΜΜΕ είναι αλήθεια ότι ασχολήθηκαν πολύ με το θέμα και από ό,τι φαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα αναθεωρήσει τα, αυτά τα σχετικά εθνικά άνω όρια Και τα αν αναρωτιούνται τι θα γίνει όσον αφορά με τη σχετική οδηγία, με τη μετανότατα όρια εκπομπών. Ε, αυτό είναι το βασικό θέμα, οπότε επιφυλάζομαι να απαντήσω σε ερωτήσεις αφού θα έχουν τεθεί. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Επιτροπή. Yeah. Thank you very much, Mr. Chairman, and um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τα αξιότιμα μέλη για την ερώτηση, παρόλο που δεν είναι εδώ τώρα. Βεβαιώνω την, Επιτροπή εξ ονόματος της Κομισιόν ότι η Κομισιόν γνωρίζει πολύ ε, καλά τα ε, θέματα αυτά της ποιότητας ε, της ατμόσφαιρας, ε, όζων, οξύδια του αζότου και άλλα εμείς γνωρίζουμε επίσης στην Κομισιόν ότι οι ρηπαντές υπολογίζεται ότι στοιχίζουν, ε, ε, μας κοστίζουν περίπου μισό εκατομμύριο πρόωρους θανάτους και σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον μέσω της οξύνησης, του ευτροφισμού και της μείωσης του όζοντος. Ανεξάρτητα από τα ΜΜΕ, θα ήθελα να σημειώσω ότι η Κομισιόν ε, τηρεί τη δέσμευση που έχει αναλάβει για αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών για την ατμόσφαιρα και ε, ενίσχυση τους όπου χρειάζεται για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Θα συνεχίσει με στοχευμένες προσεκτικά δράσεις σε διάφορα μέτωπα. Η αναθεώρηση της σχετικής οδηγίας για τα νότατα όρια πράγματι ανεβλήθη από το 2007 για να μπορέσουμε να εγκρίνουμε ένα πρόγραμμα για το κλίμα το οποίο ε, ήταν ε, αναμενόμενο να δώσει ποιοτικά ωφέλη. Το μεταξύ σημειώθηκε πρόοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους περισσότερους ρηπαντές προβλέφθηκαν μειώσεις για το 2010. Αυτά τα όρια θα τηρηθούν και αυτό είναι καλό για το διοξίδιο του θείου, την αμμονία. Τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα από, ε, από το στόχο και για τις ε, οργανικές πληθυντικές ενώσεις είμαστε στο, στόχο μας. Αυτό ισχύει και για τα οξύδια του αζότου ως ένα βαθμό που φαίνεται ότι ξεφεύγουμε κατά 10% από το στόχο. Όμως η εικόνα είναι λιγότερο θετική όταν πάμε στην κατάσταση αναχώρα. Διάφορα κράτη-μέλη ε, ήθελα, ε, ε, έχουν πετύχει το στόχο και όχι μόνο στη οξύδια του αζότου. Αλλά όχι, είναι πολύ σημαντικό να τηρηθεί η οδηγία, τώρα θα πρέπει να αναθεωρηθεί. όχι μόνο ο Επίτροπος Πορτότσνικ, αλλά όλοι οι Επίτροποι. Και αυτό κατοπτρίζεται από το γεγονός ότι τις επόμενες εβδομάδες οι Επίτροποι θα συζητήσουν την αναθεώρηση της οδηγίας ε, για τα ανώτατα όρια. Ε, γι' αυτό δεν μπορώ τώρα να σας δώσω λεπτομέρειες σε σχέση με το ε, πότε ακριβώς θα γίνει η αναθεώρηση. Πάντως η συζήτηση θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Κατόπιν τούτου τονίζω ότι μία αναθεώρηση της οδηγίας, μην έχετε καμία αμφιβολία, να μην υπάρχει καμία ε, ανασφάλεια, ε, η αναθεώρηση αυτή δεν θα δώσει τα ε, καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ούτω ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας σε σχέση με τις δεσμεύσεις στα πλαίσια του έκτου περιβαλλοντικού προγράμματος πλαίσιο γιατί δεν μπορεί η οδηγία αυτή να ειδωθεί αποκομμένη. Είναι ένα ε, αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής της Ένωσης για την ποιότητα της ε, ατμόσφαιρας. Εδώ χρειάζεται ε, συμμόρφωση, ενισχυμένη δράση. τώρα έχει ασκήσει προσφυγή κατά 20 κρατών μελών οικοπισιών που έχει ζώνες ε, όπου υπάρχει υπέρβαση των ρηπαντών. Φαίνεται ότι εδώ θα προσθεθούν δυστυχώς και τα οξύδια του αζότου. η ό,τι αφορά το επίμονο πρόβλημα των ε, ε, σωματιδίων και του οξυδίου του αζότου, ε, η Κομισιόν βλέπει την ανάγκη για επιτόπια μεγαλύτερη προσπάθεια, ιδιαίτερα όταν υπάρχει αύξηση για πρόβλεπτους λόγους. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, οι δράσεις μπορεί να έχουν σχέση με εθνικά όρια εκπομπών, που διάφορα κράτη-μέλη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, και μιλώ μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ε, είναι πιθανό να, έχουν, ε, να μην έχουν πετύχει το μέγιστο ε, όριο για το 2010. Μέχρι τώρα η Επιτροπή εστίασε τις προσπάθειες σε καλά στοχευμένα μέτρα τα οποία θα συμβάλλουν στη σημαντική μείωση των εκπομπών. Για παράδειγμα, μετά από μια μακρά διαδικασία πρόσφατα χαιρετήσαμε τη σημαντική συμφωνία για ενισχυμένη οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές που θα επιτύχει μείωση των εκπομπών οξυδίων του αζότου, του θείου και των ε, σωματιδίων. Επίσης η Κομισιόν και τώρα κύριε Πρόεδρε περνάω στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Η Κομισιόν θέλει γύρω στο τέλος του χρόνου να εγκρίνει πρόταση μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο της Συμφωνίας του 2008 σε επίπεδο IMO, το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, για σημαντική μείωση του θείου από τα καύσιμα των πλοίων. Έτσι λοιπόν, οποιασδήποτε αναφορές των ε, μέσων ενημέρωσης ε, για τη συμφωνία αυτή είναι λάθος. Η Κομισιόν έχει χαιρετήσει το, την, τις νέες διατάξεις IMO Marple γιατί οι ενδείξεις ε, μας λένε ότι οι διατάξεις αυτές θα επιτρέψουν μείωση εκπομπών του, των οξυδίων του αζότου και του θείου κατά 9, 19%. Και θα έχουμε 75% μείωση, α, 90% στην πρώτη περίπτωση και 75% για τα σωματίδια. Η πρόταση μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο της συμφωνίας που ε, σε επίπεδο με τον IMO ε, θα λάβει χώρα ε, στις αρχές του έτους μαζί με μια έκθεση για την εφαρμογή της τωρινής οδηγίας για το θείο. Η έκθεση θα περιλαμβάνει ε, δεδομένα για την σχέση κόστους-οφέλους, και ε, επέκταση των ε, περιοχών ελέγχου ε, πέρα από τις υπάρχουσες στο Τιμάνχη, τη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα. Η Κομισιόν δεν είναι μέρος συμβαλόμενο στην ΑΕΜΟ, έτσι λοιπόν δεν μπορεί να κάνει τίποτε περισσότερο από το να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη που είναι συμβαλόμενο στον ΑΕΜΟ να ζητήσουν νέες οίκας για το θείο, περιοχές ελέγχου δηλαδή, για το θείο και για το άζωτο ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μετά θα συνεχίσουμε με περαιτέρω τροπολογίες για να συμπεριλάβουμε νέες οίκα και νίκα. Ε, σε το χρόνο και αυτό θα γίνει περίπου το 2013 όταν θα ολοκληρώσουμε την ε, επανεξέταση των πολιτικών της Ένωσης. Με αυτές τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι μπορέσαμε να ασχοληθούμε και να καταπιαστούμε με το πρόβλημα και τις ανησυχίες που θέτουν τα ε, οι αξιότιμοι βουλευτές. Συντάκτες, δεν είναι εδώ, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν ικανοποιημένοι με τις απαντήσεις σας. Κρίστε, μια στιγμή να σου δίνω λίγο χρόνο να πιω στο νερό σου για να μιλήσω κι εγώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις απαντήσεις και ξεκαθαρίστε κάποια από τα σκοτεινά σημεία. Υπάρχει μεγάλη πίεση που δημιουργήθηκε λόγω των ε, δημοσιευμάτων του τύπου. Ε, ο Επίτροπος Ποτόσνικ ε, μας έδωσε την ιδέα ότι δεν θα υπάρξει τέτοια αναθεώρηση τη οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια. Επίσης, συμφωνώ και γνωρίζω ότι η Κομισιόν δεν είναι συμβαλόμενο μέρος. Αλλά όταν δίνετε, στέλνετε τέτοια μηνύματα, ε, σημάδια στα κράτη-μέλη, νομίζω ότι θα πρέπει παράλληλα να του δίνετε και σημάδι για το κατά πόσο θα πρέπει να εφαρμόσουν και τι ανώτατε τιμέ. Θα πρέπει η Κομισιόν ότι τα νέα αυστηρότατα όρια, αυστηρότερα όρια για το θείο ε, του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας θα πρέπει να εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο γιατί είναι πολύ σημαντικά για την αναθεώρηση της οδηγίας για τις άνωτες ε, τιμές εκπομπών. Καλό είναι που συζητήθηκαν ευρύτερα στην Κομισιόν είναι σημαντικό όμως, τονίζω, να γίνει αναθεώρηση, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να ετοιμάσουμε ανώτατε τιμέ για τη σωματιδιακή ύλη 2,5. Επίσης, για το θείο. Εδώ και χρόνια δεν έχουμε ε, νέα νομοθεσία. Και είναι σημαντικό ε, να αναθεωρήσουμε και το θέμα της σωματιδιακής ύλης. Χαίρομαι που θα συζητηθεί λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας υποστηρίζουμε στο Κοινοβούλιο και ελπίζω να προκύψει στα τέλη του έτους μια καλή αναθεώρηση για τα, για τα ανώτατα όρια εκπομπών. Κρίστεν, θες να ξαναπάρεις το λόγο? Καλύτερα θα ήταν να είχαμε θέσει αυτό το ερώτημα στον Επίτροπο παρά Στου υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν συζητήσαμε πρώτη φορά την ε, οδηγία για τα ανώτατα όρια, τα επιχειρήματα ήταν πολύ σαφή. Ότι σώζουμε ανθρώπινε ζωές, αν έχουμε τέτοια πρότυπα, και υπάρχουν και οικονομικά ωφέλη. Γιατί γίνονται λιγότερε ζημίες στις ε, σοδιές κτλ. Αλλά νομίζω η διάθεση για περιβαλλοντική βελτίωση σε αυτούς τους τομείς ε, δεν υπάρχει στην Κομισιόν. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν έχει εμπιστοσύνη πια στις συστάσεις των ε, συμβούλων της. Υπάρχουν πολύ σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά ωφέλη από αυτές τις βελτιώσεις. Δεν έχετε τη θέληση, Κομισιόν, να αντιμετωπίσετε τις ε, δίστροπες κυβερνήσεις που δεν θέλουν να εφαρμόσουν τα αυστηρότερα πρότυπα ή να αυξηθούν αυτές οι τιμές. Να γίνουν δηλαδή πιο αυστηρές. Δεν είναι θέμα μόνο βελτίωσης του περιβάλλοντος. Απλώ υπάρχει προθυμία στα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν την Κομισιόν. Ε, για μια πιο φιλόδοξη αναθεώρηση οδηγίας. Yes, of course, you will have the floor again. Να δώσω το λόγο, Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν δύο τμήματα στη συζήτηση να τα ξεχωρίσουμε. Για το περιεχόμενο σε θείο των καυσίμων, επαναλαμβάνω ότι ο το περιεχόμενο του θείου στα καύσιμα, η πρόταση μεταφοράς ε, του παρατήματος 6 του Διεθνούς ε, Ναυτιλιακού Οργανισμού, η ένταξη λοιπόν θα γίνει στο τέλος του έτους. Το δεύτερο θέμα είναι τα επιπλέον νίκα και σίκα ε, για τα, όσον αφορά τα ανώτατα όρια. Εδώ τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν προτάσεις στον IMO. Ε, υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη προς αυτή την κατεύθυνση. Τα νέα πρότυπα στα καύσιμα θα μεταφερθούν όμως και θα εφαρμοστούν στο τέλος του χρόνου. Αυτή είναι η απάντηση. Τώρα, για το άλλο τμήμα της ε, ερώτησης, για την οδηγία για τα ανώτατα όρια. Δεν ξέρω αν ο βουλευτής άκουσε όλη την απάντηση που έδωσα. Είπα. Ως απόδειξη της αποφασιστικότητας της ε, Επιτροπής σας λέω ότι πραγματικά ανασκουμπωνόμαστε εναντίον όλων των υπερβάσεων των ανωτάτων ορίων στα κρατη Το εξήγησα. Εξήγησα γιατί ε, αναβλήθηκε η αναθεώρηση. Για να επιτρέψουμε στο πακέτο κλίματος και ενέργειας να περάσει, ούτως ώστε να υπάρξει πραγματική βελτίωση στην ποιότητα του αέρα. Και μετά από αυτό, είπαμε, θα ξανακάνουμε τους υπολογισμούς σε τεχνικό επίπεδο και ο Επίτροπος Ποτότσνικ συζητάει μαζί με τους υπόλοιπους επιτρόπους, το σώμα των επιτρόπων, για το ποια είναι η καλύτερη στιγμή για να τα προτείνει αυτά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι από μόνη της αυτή η οδηγία για τα ανώτατα όρια εκπομπών δεν πρόκειται να μας δώσει τα ωφέλη που περιμένουμε. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν αυτά τα εθνικά ανώτατα όρια σε ό,τι αφορά τις διεθνείς κινήσεις ε, πλοίων και τη μόλιση που υπάρχει, αλλά και η τοπική δράση είναι σημαντική. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά τα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν εκ του σύνεγγης. Για το σχόλιο τώρα που έκανε ο βουλευτής για τη σημασία ύπαρξης νομοθεσίας για τη σωματιδιακή ύλη, επίσης συμφωνώ. Έχετε απόλυτο δίκιο, τι να σας πω. Αυτά προς το παρόν. I'm, σίγουρα ε, πρέπει να έρθουν τα μέτρα γιατί υπάρχει μεγάλη ανάγκη και πολλοί κόσμος Το ε, Επόμενο θέμα τώρα είναι το υπαρισμό 7 και αυτό αφορά την αναθεώρηση τη οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη από τους που συμπέραγαν ποιο ε, Κρήτονα. Θε να λάβει εσύ το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μετά τη θεομηνία στο Μεξικό αυτού του ατυχήματο, όλοι συνειδητοποίησαμε τι προβλήματα, τι κενά υπάρχουν ε, στην ε, νομοθεσία τη δική μας αλλά και γενικότερα και όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου, πρεσμό του κινδύνου αλλά και όσον αφορά τον επιμερισμό της ευθύνης για ε, όλα όσα έγιναν στον κόλπο του Μεξικού, την έκρηξη και αυτά στην αρχή. Βεβαίω είχαμε την εξόρυξη του πετρελαίου, επίσης όμως είχαμε και το μεθάνιο, το οποίο ε, ξέφυγε κάνουμε τις διαρροής και είπαμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά την θάλασσα. Διαπιστώσαμε ότι οι υπολογισμοί μας έχουν πάρα πολλούς περιορισμούς όσον αφορά την του <clears throat> Το μεθάνιο είναι αέριο και υπάρχει και ένα άλλο αέριο το οποίο χρησιμοποιούμε. Ε, έχουμε, έχουμε το CCS όσον αφορά δηλαδή τη δεξαμενή απορρόφηση και την ε, αποθήκευση του διοξιδίου. Ε, είχαμε κάνει διάφορα, αλλά παρόλα αυτά δεν ήμασταν όπως έπρεπε προετοιμασμένοι και από ό,τι φαίνεται χρειάζεται να αναβαθμίσουμε, να ενισχύσουμε, να βελτιώσουμε την οδηγία αυτή για κάθε ενδεχόμενο. Ιδίω να δούμε τι θα ισχύσει άπαξ και αυτή η οδηγία δεν καλύπτει ατυχήματα στην ανοιχτή θάλασσα και όσον αφορά εργασίες γεώτρησης. Άρα, αν θεωρηθεί η οδηγία πνευματική ευθύνη και επομένω να καθιερωθεί αυστηρή ευθύνη για κάθε είδου εργασίες γεώτρηση, εξόριξη, έγχυση, και σε ανοιχτή θάλασσα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και επ' αυτού περιμένω να ακούσω τη γνώμη τη ε, Επιτροπή να μα εξηγήσουν τι πρωτοβουλίε θα αναλάβουν για την ευθύνη που προκύπτει από αυτέ όλε τι εργασίε, έγχυση, γεώτρε κλπ. Δεν βλέπω κάποιο άλλο να θέλει υποβάλει ερώτηση, επομένως θα δώσω τα δυστυχία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιο είναι, ο κύριος Γκαρθία. Α, μάλιστα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Κομισιόν ήδη ανακοίνωσε στην Ολομέλεια του Ιουλίου ότι μετά το ατύχημα αυτό θα άρχιζε μια διαδικασία με διπλό στόχο. Πρώτον, εντοπισμό πιθανών κενών στην υφισταμένη νομοθεσία της Ένωσης και δεύτερον, για να καθοριστεί αν νομοθετική δράση χρειάζεται ενδεχομένως για την πλήρωση αυτών των κενών. Η αξιολόγηση αυτή ακόμα συνεχίζεται, αλλά κάποια προκαταρκτικά δεδομένα αρχίζουν να διαφαίνονται σε ό,τι αφορά την οδηγία περιβαλλοντικής ε, ευθύνης. Το πρώτο πόρισμα είναι ότι η γεώτρηση πετρελαίου στην ανοιχτή θάλασσα καλύπτεται από την οδηγία περιβαλλοντικής ευθύνης και σε αυστηρό καθεστώς ευθύνης. Η εξόρυξη πετρελαίου σε ανοιχτή θάλασσα είναι μια επαγγελματική δραστηριότητα η οποία συνεπάγεται χειρισμό επικίνδυνων ουσιών και το πετρέλαιο το ίδιο είναι επικίνδυνη ουσία, ορίζεται ως τέτοια και ο χειρισμός, διαχείριση επικίνδυνων ουσιών είναι μια δραστηριότητα που αναφέρεται στο παράρτημα 3 της οδηγίας. Δεύτερον, οι αναλύσεις μας δείχνουν ότι η προστασία ειδών, θαλασσίων ειδών, ε, αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής. Στα θαλάσσια ύδατα καλύπτονται οι φυσικές καταστροφές σε ύδατα ε, στο οποίο έχει αρμοδιότητα το παράκτιο κράτος. Ιδιαίτερα εδώ περιλαμβάνονται τα χωρικά ύδατα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η οδηγία αυτή περιβαλλοντικής ευθύνης όμως θα πρέπει να καλύψει είδη τα οποία προστατεύονται από ενωσιακό δίκαιο ή και εθνικό δίκαιο εάν τα κράτη-μέλη επιλέξουν αυτή τη λύση. Δηλαδή η ζημία στα εμπορικά θαλάσσια είδη δεν καλύπτεται από την οδηγία περιβαλλοντικής ευθύνης. Αυτό είναι οικονομική ζημία εν προκειμένου η οποία καθ' αυτή δεν καλύπτεται από την οδηγία σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη. Έπειτα, ο... ένας τομέας όπου υπάρχει σαφές κενό στην κάλυψη της οδηγίας περιβαλλοντικής ευθύνης αφορά την ε, καταστροφή των υδάτων. Εδώ είναι μερική η κάλυψη από την ε, Οδηγία Περιβαλλοντικής Ευθύνης, δηλαδή ε, η βλάβη οικολογικής ποιότητας καλύπτει μόνο τα παράκτια ύδατα, όχι πέραν του ενός ναυτικού μιλίου και η ζημία στη χημική σύνθεση των υδάτων καλύπτεται αλλά όχι ικανοποιητικά. Και δεν ξεπερνά τα χωρικά ύδατα. Η ζημία στα ύδατα, στην φαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη δεν καλύπτεται από την οδηγία περιβαλλοντικής ευθύνης. Ε, φαίνεται ότι το κενό αυτό στο γεωγραφικό εύρος εφαρμογής της οδηγίας στα θαλάσσια ύδατα θα πρέπει να καλυφθεί. Καταρχήν αυτό θα απαιτήσει τροπολογία στην οδηγία περιβαλλοντικής ευθύνης, ούτως ώστε η τελευταία να ευθυγραμμιστεί με νεότερη ε, ενωσιακή νομοθεσία δηλαδή την Οδηγία Στρατηγικής Θαλασσίου Περιβάλλοντος. Τώρα, ίσως διαφορά το δεύτερο θέμα που ετέθη στην προφορική ερώτηση, ευθύνη και δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, εκεί κατά τη γνώμη μας δεν υπάρχει κενό στην κάλυψη του θέματος από την Οδηγία Περιβαλλοντικής Ευθύνης. Λειτουργία σημείων αποθήκευσης ε, σύμφωνα με την Οδηγία Δέσμευσης και Επαγίδευσης του Άνθρακα αποτελεί μία από τις δραστηριότητες που απαριθμείται στο παράρτημα 3 της Οδηγίας Περιβαλλοντικής Ευθύνης και το μόνο πρόβλημα που εντοπίζουμε σε αυτό τον τομέα αφορά ίσως τη δυσκολία που υπάρχει για να γίνει μια σωστή αξιολόγηση της ζημίας. Θα έλεγα όμως ότι το πρόβλημα αυτό δεν αποκλειστικά αυτόν τον τομέα, απαντάται και σε άλλου είδους ζημίες που οφείλονται σε άλλου είδους δραστηριότητες. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό το μεθοδολογικό πρόβλημα δεν είναι καθ' αυτό ανυπέρβλητο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ σαφής νομίζω η απάντηση. Κρήτον, ε, θέλεις ζητήσει το λόγο πάλι. Εκτός μικροφώνου κύριος Αρσένης. Όπως θέλει μπορεί να μιλήσει πρώτος. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απάντησή της. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν κενά παρόλα αυτά. Ανάλογα με αυτά που υπάρχουν ε, στην νομοθεσία για την εξόριξη πετρελαίου. Το βασικό είναι ότι η Κομισιόν έχει διάθεση να αναθεωρήσει την οδηγία. Θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγι τι προτάσεις τη για να βεβαιωθούμε ότι αυτή τη φορά θα καλύψουμε τα κενά και θα αποφύγουμε την, τις πετρελαιοκυλίδες και τις όποιες καταστροφές στα υδατά μας. Ο Μπάζ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά από αυτά που είπε ο Κρήτον, Αρσένης, θέλω να ξεκαθαρίσουμε το εξή. Φυσικά, ευχαριστώ την Επιτροπή για τις απαντήσεις. Κατάλαβα τώρα πού υπάρχουν τα κενά, μια ιδέα μπασχετός τα κενά στην οδηγία υπάρχουν δύο βασικά κενά. Ε, γεωγραφικά κενά, μιλάμε για τα νερά, δηλαδή τι χημική βλάβη και μόλις υπάρχει στο είδωρ. Δεν μιλάμε γενικά για το είδωρο σε όλη την Ευρώπη. Ε, δεν καλύπτεται όλο το νερό από την οδηγία για την ευθύνη και το άλλο είναι ε, το γεγονός ότι κάποια είδη, παραδείγματος χάρη εμπορική αλία, δεν καλύπτεται. Δηλαδή, όταν η Κομισιόν τελικά θα κάνει την ανάλυση της θα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για να τροποποιήσει την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη, ούτω ώστε αυτά τα δύο κενά να καλυφθούν για το τη γεωγραφική κάλυψη και για τα είδη. Θα σα ξαναδώ στο λόγο Κομισιόν. Επιπλέον, πότε θα έχετε Κομισιόν τα τελικά συμπεράσματα, πότε θα μα τάσει η πρόταση και δεδομένε τη περιπλοκότητα για το ποιο έχει την ευθύνη, ποιο έχει την ιδιοκτησία, ποιος δραστηριοποιείται. Η οδηγία για την ευθύνη, την περιβαλλοντική ευθύνη ξεκαθαρίζει τον επιμερισμό των ευθυνών. Η έλλειψη κάλυψης των εμπορικών ειδών από την Οδηγία για την Περιβαλλοντική Ευθύνη δεν συνιστά κενό του συστήματος αυτό καθεαυτό. Η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη σχεδιάστηκε ειδικά για να καλύψει την περιβαλλοντική ζημία. Αυτό που λέτε εσείς είναι κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική βλάβη, μια διαφορετική ζημία. οικονομικής φύσεως κυρίως και νομίζω απαιτεί διαφορετικό μέσο. Όχι αυτή την οδηγία περιβαλλοντικής ευθύνης. Για το δεύτερο ερώτημα. αν θα σας υποβληθεί ένα σχέδιο με σκοπό την τροποποίηση της οδηγίας περιβαλλοντικής ευθύνης. Τις επόμενες μέρες θα υποβάλουμε μία έκθεση για την οδηγία της, ε, για την εφαρμογή της οδηγίας περιβαλλοντικής ευθύνης. Και θα μιλήσουμε όλος ιδιαίτερο για το κατά πόσον υπάρχουν μηχανισμοί οικονομικοί μηχανισμοί και θα αναφερθούμε και στις α, τροπολογίες που πρέπει να γίνουν σε αυτή την οδηγία, ούτως ώστε να υπάρχει η σωστή και πλήρης κάλυψη των ζημίων που προέρχονται από τις ε, δραστηριότητες εξόριξης ε, πετρελαίου στις πλατφόρμες. Η πρόταση όμως ήταν τμήμα ενός ευρύτερου πακέτου προτάσεων. Ούτως ώστε να υπάρχει πλήρη κάλυψη της γεώτρησης ε, πετρελαίου από τις πλατφόρμες. Η οδηγία περιβαλλοντικής ευθύνης είναι ένα τμήμα, μια ψηφίδα του πακέτου. Υπάρχουν και άλλες πτυχές που είναι σημαντικές και ίσως πρέπει να αναλυφθεί δράση. Ευχαριστώ. Και ένα τελευταίο για το χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, για πόσους μήνες μιλάμε από τώρα. Α, δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα σε αυτό το στάδιο γιατί υπάρχουν πολλές γενικές διευθύνσεις, ε, συμμετέχουν πολλοί επίτροποι, πάντως γίνεται μια πολύ δραστήρια δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Δυστυχώς πάντως δεν είναι δυνατόν σε αυτό το στάδιο των εργασιών να πούμε κάτι περισσότερο σε σχέση με το πότε θα κατατεθούν οι προτάσεις. Θα κατατεθούν το συντομότερο. Α, δηλαδή θα δράσετε γρήγορα για να μην κάνουμε κι άλλη προφορική ερώτηση πάνω στο θέμα πριν ε, αναλάβετε δράση. Αν κατάλαβα καλά την Κομισιόν, όταν είναι εμπορικά τα είδη, δεν καλύπτονται από την ΕΛΔ, την Οδηγία Περιβαλλοντικής Ευθύνης, γιατί δεν θεωρούνται δηλαδή περιβαλλοντικά είδη τα είδη. Δηλαδή πώς θα το εξηγήσουμε αυτό στους αλληλείς. Αν πάθουν ζημιά τα ψάρια και δεν μπορούν να τα πιάνουν οι αλληλείς, πού θα καλύπτεται η ζημία. Αν δεν καλύπτεται από την οδηγία περιβαλλοντική ευθύνης και λέτε δεν είναι κενό αυτό, ε, τότε πού καλύπτεται. Γιατί σε τελευταία ανάλυση η ζημιά που παθαίνουν τα ίδια αυτά πρέπει και αυτή να καλύπτεται από τις εταιρείε που ρισκάρουν, αν θέλετε, την εξόριξη πετρελαίου. Να το εξειδικεύσετε αυτό, γιατί αν δεν εμπίπτει στην οδηγία περιβαλλοντική ευθύνη, τότε πού εμπίπτει. Μάλιστα. Κομισιόν. Ευχαριστώ. Προς το παρόν αυτές οι ζημίες καλύπτονται από αστική ευθύνη, καθεστώτα αστικής ευθύνης που έχουμε αναπτύξει σε όλα τα κράτη-μέλη. Εκεί υπάρχει σαφής κάλυψη περιπτώσεων βλάβης, ζημίας στους αλληλείς ή σε οποιαδήποτε άλλη ε, οικονομική δραστηριότητα, τουρισμό, ακόμα και ζημία στην ιδιοκτησία. Η οδηγία περιβαλλοντικής ευθύνης αρχικά ευθύς εξ αρχής σχεδιάστηκε ως προσπάθεια να καλυφθεί το κενό που υπήρχε εκείνη, εκείνη την εποχή. Η περιβαλλοντική ζημία δεν είναι οικονομική ζημία, άρα δεν καλύπτεται από τα καθεστώτα αστικής ευθύνης και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι υπήρχε ανάγκη να εγκριθεί αυτό το ειδικό μέσον για την περιβαλλοντική ευθύνη. Ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη ερώτηση, που είναι εντελώς διαφορετικό θέμα. Βέβαια έχει επίδραση στα ζώα. Υγειονομικοί κανόνες για τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Ποιον έχουμε εδώ, Χρήσε, εσύ έκανες μεταξύ άλλων την ερώτηση. Θέλεις να λάβεις το λόγο λοιπόν εσύ. Να ακούσω την απάντηση και να επανέλθω. Έχω διάφορα ονόματα εδώ. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν που θα απαντήσει, ας μας πει και το όνομά του παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Αλμπέρτο Λαντόμαντα και είμαι επικεφαλής της ε, ε, μονάδας ε, για την υγεία των ζώων στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας των ζώων, της υγείας των ζώων. Χαίρομαι για την ευκαιρία που μου δίνετε να ενημερώσω για, τα, για το φάκελο ζωικών υποπροϊόντων. Πέρσι ο κανονισμός 1069 του 2009 εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αυτό το νομοθέτημα εισάγει πιο αναλογικές, αναλογικούς υγειονομικούς κανόνες για τα ισοϊκά προϊόντα που δεν καταναλώνται τον άνθρωπο. Και αυτός ο κανονισμός καλύπτει πάρα πολλά υλικά εκτός της διατροφικής αλυσίδας για, την, για, για κτηνοτροφές ή για ε, λιπάσματα ή για άλλου είδους τεχνικά προϊόντα. Αίμα, δέρμα για μέσα διάγνωση στα εργαστήρια. Ο δε κανονισμός προσδίδει αρμοδιότητε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημαντικέ, ώστε να εφαρμόσει τεχνικέ λεπτομέρειε όπω τα, τα, τα, πρότυπα υγιεινή, ε, την επεξεργασία και άλλε προποθέσει και ε, ε, έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις που έχει τάξει ο νομοθέτης, οπότε άρχισε τις διαβουλεύσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους εμπλεκόμενους, με τα κράτη-μέλη και με τρίτες χώρες, που η βασική μας εμπορική εταίρεια και πρόκειται επομένω περί μέτρων οικονομικά σημαντικών, οπότε σε αυτή την φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκληρώνει τα προτινόμενα μέτρα για να υλοποιηθεί ο βασικός κανονισμός. Και στη συνέχεια θα υποβληθούν όλα αυτά ή στην ε, μόνιμη επιτροπή τον επόμενο μήνα που ασχολείται με τα θέματα υγείας διατροφής και σύμφωνα με την πράκτη προβόμενη διαδικασία για τον κανονιστικό έλεγχο θα υπάρχει δυνατότητα αναθεώρησης ε, στο μέλλον λεπτομερέστερης. Παρ' όλα αυτά, με μεγάλη μου χαρά, ε, που σας ενημερώνω σε το πώς έχει σήμερα κατάσταση των πραγμάτων όσον αφορά τα προτινόμενα μας μέτρα. Όσον αφορά τους εφαρμοστικούς κανόνες, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε ε, στα όσα εσάς σας προβλημάτισαν ως εξή. Απλούστεροι κανόνες και έτσι θα έχουμε 30 χωριστά μέτρα τα οποία είχαν προβληθεί στις προηγούμενες διατάξεις αλλά τώρα θα έχουμε μια κωδικοποιημένη ενιαία ε, νομοθετική πρόταση τώρα όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία παίρνουν από μεταποίηση θα δούμε πώς θα έχουμε ορίσει ένα συγκεκριμένο σημείο ελέγχου ε, στην, στην, ε, στην, στην ε, όσον αφορά το, το biodiesel, όσον αφορά τροφές για κατοικίδια και με διάφορες μεθόδους μεταποίησης, τόσο ώστε να είναι δυνατόν τα υλικά να καθαρίζονται αυτά που αφορούν ιατρικές διαγνώσεις και έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία με τη νέα νομοθεσία, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει ανιχνευσιμότητα και έτσι θα υπάρχει το περιθώριο για αναλογικούς ελέγχους όσον αφορά τα εργαστήρια που αναλύουν τα προϊόντα από εγκαταστάσεις μετα, μεταποίησης και το λεγόμενο κομποστάζ. Και έτσι έχουμε αυτόν τον κανονισμό βάσης όσον αφορά το ποια προϊόντα καλύπτονται από αυτήν την νομοθεσία για την υγεία των ειδών διατροφής. Η έλεγχη επομένω θα είναι πιο αναλογική. Θα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με το πώ μπορούμε να πετύχουμε κάποιου στόχου, ιδίω όσον αφορά τα μέσα μεταφορά για διάφορε. Διάφορες Διαφορετικές διαφορετικά προϊόντα, τα οποία όμως παράγονται Στι ίδιε εγκαταστάσει, στο ίδιο εργοστάσιο. Στον αφορά τα παραπροϊόντα, ε, τα, ζωικά, θα πρέπει να διέπονται από την ομοθεσία που προστατεύει τη και άρα θα πρέπει να υπάρχει ομοιογενής προστασία παντού προς όφελος των Ευρωπαίων. Αυτές είναι οι προθέσεις μας, τους δε πρόσφατους τελευταίους μήνες. Έχουμε συνεχή επαφή με τον κύριο Σνέλχαρ που ήταν ο εισηγητής του κανονισμού 1069 του 9 και η συνεργασία ήταν πάρα πολύ θετική. Τον ευχαριστούμε και τώρα με χαρά να ακούσουμε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής σας όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που αναλάβαμε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και τώρα ο κύριος Σύνχαλα Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ την Κομισιόν γιατί είχαμε μια ευχάριστη συνεργασία και καταφέραμε ένα σύνθετο ντοσιέ να το εγκρίνουμε σε πρώτη ανάγνωση. Αυτό εδράζεται στην καλή συνεργασία με την Κομισιόν και με την Τσεχική Προεδρία τότε. Θέλαμε, πριν εγκριθεί ο εφαρμοστικός κανονισμός τότε, να γίνει μια παρουσίαση εδώ στην Επιτροπή. Έγινε αυτό τώρα και νομίζω ότι η Κομισιόν και εδώ κτήρισε το λόγο της. Γενική παρατήρηση για τον φάκελο αυτό. Πάντα τρομάζω όταν εγκρίνουμε κανονισμούς που καλύπτουν ε, ένα συγκεκριμένο τομέα και μετά ε, έρχονται οι συγκεκριμένοι εφαρμοστικοί κανόνες ε, που μπορεί να μην τα καλύπτουν όλα ή που ε, δημιουργούν και γραφειοκρατικά εμπόδια. Δεν είναι ο στόχος μας βέβαια η μείωση της γραφειοκρατίας. Είναι γραφειοκρατική η ζούγκλα που αντιμετωπίσαμε και που πρέπει να συζητήσουμε γενικότερα. Και να δούμε αν χρειάζονται όλοι αυτοί οι πολύ και λεπτομερείς κανόνες. Αυτό το λέω ε, αυτή τη στιγμή εν παρόδο, αλλά ως βάση μιας μελλοντικής συζήτησης. Λοιπόν, ήρθε το έγγραφο, έχουμε χρόνο να αποφανθούμε και να το σχολιάσουμε. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε ορισμένα πράγματα που αποτελούσαν τους στόχους που είχαμε, θέλαμε, γιατί θέλαμε ένα νέο κανονισμό γιατί υπήρχαν οι κανονισμοί υγειονομικοί, εδώ δεν υπήρχε συμφωνία. Θέλαμε να συμφωνήσουμε και να έχουμε μία ξεκάθαρη βάση για τα ζωικά υποπροϊόντα. Ε, θέλαμε διατάξεις, αυτή ήταν μια μεγάλη επιθυμία από, τους βόρειους, ε, από τις βόρειες χώρες, σκανδιναβικές χώρες, να ρυθμιστούν τα ζωικά υποπροϊόντα και Μα ενδιέφερε να διασφαλίσουμε την ειχνηλασιμότητα ή ανιχνευσιμότητα και να διασφαλίσουμε την προστασία των καταναλωτών από αυτά τα προϊόντα. Οι στόχοι που γράψαμε τότε και στον κανονισμό, στον ε, παρόντα κανονισμό έχουν συμπεριληφθεί όλα με ωραίο τρόπο. Πολλά ζητήματα που συζητήσαμε τότε έχουν σαφώς εντοπιστεί ε, για το end point, το τελικό σημείο ορίζεται πολύ ξεκάθαρα πότε είναι τελικό το σημείο, δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο. Βέβαια θα πρέπει να καταπιαστούμε πιο εντατικά με το θέμα αυτό. Αλλά εν πολλής, ε, τώρα εγώ είμαι ικανοποιημένο. Τώρα για το ε, προϊόντα είχαμε αναθέσει στην Κομισιόν μαζί με το Συμβούλιο και με την ΕΦΣΑ που θα γνωμοδοτούσε και πρέπει να δουλεύει πιο γρήγορα η ΕΦΣΑ γιατί εγώ περίμενα αυτό το end point να αναφέρεται στον εφαρμοστικό κανονισμό γιατί διευκολύνεται έτσι η εργασία των βιομηχανιών. Τώρα, η διατροφή μικρών ζώων ρυθμίζεται καλά. Έχουμε στοιχεία για τα μικρές ποσότητες ζωικών υποπροϊόντων, 500, 500 κιλά αναφέρεται. Πώς ελέγχονται αυτές οι ποσότητες, ε? πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε. 50, 50, 50 χιλιόγραμμα την εβδομάδα αναφέρεται. Ε, σε ορισμέ πότε θα αρχίσουμε να μετράμε την εβδομάδα. αρχίζουν, ή σε μερικούς αρχίζει η σε μερικους αρχιζει η εβδομάδα να μετράει την Τετάρτη. Υπάρχουν ορισμένες γενικολογίες. Αλλά θα πρέπει να δούμε στην πορεία πώς θα διαμορφωθεί ο έλεγχος. Για τα διαγνωστικά θέματα είναι καλή η διατύπωση για να ε, με το endpoint, είναι πολύ εντάξει αυτά. Για τις εγκαταστάσεις βιοαερίων έχω κάποια αβεβαιότητα, αλλά δεν ξέρω, ίσως να μας το ξαναπεί η Κομισιόν. Αν θυμάμαι καλά, είχαμε αποφασίσει τότε ότι θα μπορούμε τα απορρίμματα από τις εγκαταστάσεις βιοαερίου να πηγαίνουν στους αγρούς. Δεν το βλέπω αυτό να το λέει τώρα. Εν σε η Κομισιόν στον εφαρμοστικό κανονισμό ανταποκρίθηκε καλά στις επιθυμίες μας και ε, όλα αυτά που είχαμε πει τα ε, εξέτασε, τα αξιολόγησε και τα ενσωμάτωσε και οι γνωμοδοτήσεις των, από τους εμπλεκομένους είναι θετικές ως τώρα. Οπότε όλοι νομίζω ότι ε, προχωρήσαμε ε, στην μείωση της γραφειοκρατίας, διασφάλιση της ε, υγείας και διαμόρφωση ενός τελικού σημείου end point. Νομίζω, εκτός αν διαφωνούν οι συνάδελφοι, νομίζω ότι πολύ εύκολα θα προχωρήσουμε και θα εγκρίνουμε ε, την πρόταση. Ευχαριστώ. Έχει κάποιος άλλος το λόγο, λέει ο Πρόεδρος, εσείς. από τη δική μας την πλευρά, μετά τον συνάδελφο Σνέλχαρτ, θα έλεγα ότι τα περισσότερα από αυτά που είχαμε ε, ζητήσει ε, αντικατοπτρίζονται στο κείμενο. Βέβαια, δεν μειώνεται η γραφειοκρατία τώρα, ίσως στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό θέμα και η εφαρμογή όλων αυτών των ε, εγγράφων Γενικά πάντως μπορώ και εγώ να συμφωνήσω με τον προηγούμενο συνάδελφο ότι είναι καλή η προσπάθεια, είναι καλό βήμα προς την κατεύθυνση της προστασίας της υγείας των πολιτών μας και τον καθορισμό του end point, του τελικού σημείου. Ωραία. Αν δεν ζητεί άλλο το λόγο θα ήθελα εγώ να σας ρωτήσω κάτι γιατί ένας ακτιβιστής ε, υπέρ της ε, ευημερίας των ζώων ε, είχε μια ανησυχία οι αρκούδες και οι λύκοι της Βόρειας Ευρώπης ε, καλύπτονται από δηλαδή είτε σε σταθμ, θα μπορούν να ε, διατρέφονται είτε μέσα είτε έξω τους, ε, από τους σταθμούς διατροφής των ζώων, των άγριων ζώων θα μπορούν να ε, να τρέφονται και τα άγρια αυτά ζώα, λύκοι και αρκούδες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσω. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο Σνέλχαρ και την κυρία Κάλενμπαχ. Λοιπόν, λεπτομερές ταέρες απαντήσεις θα δώσω και ίσως και ο συνάδελφος Τιμ Κούμπελεχ μπορεί να ε, βοηθήσει και να απαντήσει. Τώρα, για τα endpoints. Πώς έχουν τώρα τα πράγματα. Επαναλαμβάνω, θα ορίσουμε endpoint για το biodiesel, ε, τα δέρματα και το μάρια δέψης, ε, τα ε, διατροφές μικρών ζώων, μεταποιημένα σγούνες. Ο ολαιοχημικός τομέας υπέβαλε επιστημονικά στοιχεία στην Κομισιόν και πάνω σε αυτή τη βάση η μεταποίηση θεωρείται ασφαλής σε αυτό το τομέα. Ακόμα και αν ιστεί που έχουν προσβληθεί από την πίεση, σπογκώτηση, κεφαλοπάθεια, ε, έχουν χρησιμοποιηθεί. Πριν ε, καθοριστεί το τελικό σημείο, ή το απότερο σημείο, το endpoint, η Κομισιόν ε, έκανε διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη, δημιουργήθηκε ομάδα εργασίας και θα διαβουλευτεί και με την ΕΦΣΑ. Μάλιστα ήδη ζήτησε γνωμοδότηση από την ΕΦΣΑ και η ΕΦΣΑ μα, πρόκειται στις αρχές του 2011 να υποβάλει τη γνωμοδότηση. Τώρα, ίσως ό,τι αφορά τις μικρές ποσότητες, οι ποσότητες που συζητούμε τώρα με τους εμπλεκομένους και τα κράτη-μέλη είναι 50 χιλιόγραμμα την εβδομάδα, πολύ λιγότερο από τα 500. Ίσως ό,τι αφορά την δυνατότητα ε, ε, ε όχι μόνο των αρπακτικών πτηνών αλλά και των αρκούδων και των λύκων, αυτό θα είναι δυνατόν στους σταθμούς διατροφής των ζώων, αλλά και εκτός των σταθμών αυτών. Και για το τελευταίο θέμα, παρακαλώ να απαντήσει ο συνάδελφος, γιατί νομίζω εγώ δεν απάντησα σε μια ερώτηση του κυρίου Σνέλχαρτ. Ο συνάδελφος Τίμ Κούμπελα θα απαντήσει σε μία από την ερώτηση του κυρίου Σνέλχαρτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τις εγκαταστάσεις βιοαερίου και για τις, τη χρήση καταλήπων πέψης. Αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι ποια είναι τα πρότυπα για, την, για τη μετατροπή των ε, υποπροϊόντων των εγκαταστάσεων αυτών βιοαερίου. Ε, υπάρχουν εθνικά πρότυπα σε ορισμένα κράτη-μέλη. Αν η αξιολόγηση κινδύνου μας λέει ότι η διαδικασία αυτή είναι ασφαλής, φυσικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κατάλοιπα πέψης. Από την άλλη, σε ορισμένε περιπτώσεις μην ξεχνάμε ότι αυτά τα προϊόντα είναι αντικείμενο εμπορίου μεταξύ κρατών μελών. Επομένως υπάρχουν κάποιες ανησυχίες ότι η αξιολόγηση κινδύνου ε, που γίνεται σε ένα κράτο μέλο μπορεί να συμπίπτει με αυτή που γίνεται σε ένα άλλο κράτο μέλο. Σε ό,τι αφορά για, την, για κάποια προϊόντα συγκεκριμένη προέλευση. Πάντως ε, γεγονός είναι ότι καλύπτουμε νομίζω τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων. Ο κύριο Σνέλχαρτ, ε, και εγώ τώρα δεν είμαι πολύ σίγουρο, αλλά είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα στι εγκαταστάσει βιοαερίου που θέλαμε καλό κανονισμό και τα καταφέραμε νομίζω. αλλά σε, στην οδηγία πλαίσιο είχαμε αποφασίσει ότι οι εγκαταστάσει θα δίνουν απορρίμματα. Έτσι τα λέγαμε. Οπότε είχαμε πρόβλημα. Θέλαμε να λυθεί το πρόβλημα και η πλειοψηφία συμφώνησε. Δεν σημαίνει ότι η πλειοψηφία έχει πάντα δίκιο, αλλά υπάρχει μια αντίφαση εδώ, θεωρώ. Οπότε δεν ξέρω θα, αν έχει λυθεί το θέμα σε αυτόν τον εφαρμοστικό κανονισμό. Θα έλεγα ναι μετά τη δήλωση που ακούσαμε. Αλλά καλό είναι να το επιβεβαιώσουμε άλλη μια φορά. Κομισιόν ας απαντήσει ποιος είναι καταλληλότερος και αρμοδιότερος για αυτό το θέμα. Επιλύθηκε το πρόβλημα από πλευρά μα. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι αν οποιοδήποτε λίπασμα χρησιμοποιηθεί στη γη, όχι μόνο τα κατάλοιπα πέψης, πάντα υπάρχουν περιβαλλοντικοί κανόνες που καλύπτουν τη χρήση τέτοιων λιπασμάτων. Ε, υπάρχει και το σχετικό άρθρο για την υγεία συνθήκη. Υπάρχουν κανόνες λοιπόν που αποφασίζουν ε, τι, πάει, τι μπορεί να επηρεάσει το έδαφο, τι μπορεί να επηρεάσει τα επίγεια ύδατα κτλ. Υπόγεια ύδατα. Η νομοθεσία όμως αυτή καθ' αυτή δεν παρεμποδίζει τη χρήση τέτοιων καταλήπων πέψης. Ήταν το τελευταίο σημείο στην μερίσια διάταξη σήμερα. Ακυρώνει τη συνεδρίαση των συντονιστών. Αύριο το πρωί στις 9 θα τα ξαναπούμε για πολλές σημαντικές ψηφοφορίες και νομίζω ότι ο πρόεδρος, ο Γιώργο Λάινεν, θα θέλει να είστε όλοι ακριβείς για να ξεκινήσουμε στις 9.